σχετικά πλαίσια. Εάν οι εθνικές στρατηγικές δεν υλοποιηθούν και μεταφραστούν συγκεκριμένες μεσοπρόθεσμες Μεσοπρόθεσμα σχέδια εφαρμογή που συνδέονται με επιχειρησιακά προγράμματα και ειδικέ παρεμβάσει και προγράμματα σε τοπικό επίπεδο, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση και τα σχετικά πλαίσια δεν θα μπορούσαν να έχουν πράγματα να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν. Οι εθνικέ στρατηγικέ θα πρέπει να έχουν τοπικό χαρακτήρα και θα πρέπει να λάβουν επιχειρησιακό χαρακτήρα και τα διεθνή σχέδια θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένους στόχους, δείκτες και θα γίνεται σωστή παρακολούθηση και εποπτεία. Και σχετικά πλαίσια να Η UNDP μπορεί να βοηθήσει να δημιουργηθεί το δυναμικό για τοπική αλλαγή και για να υλοποιηθούν αυτά που θέλουμε. Το κάνουμε αυτό ποικιλοτρόπω. Εργαζόμαστε με του θεσμού σε τοπικό επίπεδο για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού όσον αφορά το τι έχει να αντιμετωπίσει ο πληθυσμό των Ρωμά. Εφαρμόζουμε αναπτυξιακά προγράμματα επί επίπεδου. Κάνουμε παρεμβάσεις σε τομείς που έχουν μεγάλο ποσοστό Ρωμά. Βοηθούμε στο να εφαρμοστούν επιχειρησιακά στρατηγικές. Μισό λεπτό κυρία Σουλτάνο Γλουλίου Πρόεδρος. Ίσως έπρεπε να σας πω πριν ξεκινήσουμε ότι έχουμε τουλάχιστον έξι ομιλητές που περιμένουν και Έχουμε και ψηφοφορία που προβλέπεται στις 12. Και πρέπει να ψηφίσουμε. Πρέπει να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα. Διότι πολλά μέλη ε, έχουν προγραμματίσει εργασίες του να έρθουν ακριβώ εκείνη τη στιγμή. Σα εκλυπαρώ, λάβετε το υπόψη για να μπορέσετε να συνοψίσετε, να είστε πιο σύντομοι. Και για τα υπόλοιπα μέλη που τώρα είναι έτοιμα να πάρουν το λόγο, τα εκλυπαρώ και αυτά να μιλήσω μόνο για πέντε λεπτά ο καθένα. Ευχαριστώ, λέει κύριε Πρόεδρε. Τελείωσα, ξεμπέρδευσα, ξεμπέρδευσα. Ε, δίγα λεπτά έχω ακόμα. Ίσως μπορώ απλώς να συνοψίσω. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι να δείξουμε ότι είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές, να προτείνουμε πώς μπορεί να επιτευχθεί αλλαγή και να πούμε ότι θα υπάρχουν πολλά ωφέλη, τεράστια ωφέλη από την ένταξη των Ρωμά όσον αφορά την ανθρώπινη εξέλιξη. Άρα σωστό δρόμο ακολουθούμε και όταν λέμε εμείς, όλοι μας δηλαδή, και είμαι σίγουρη ότι σε λίγα χρόνια στο μέλλον θα μπορούμε να κοιτάμε στο παρελθόν υπερήφανοι για αυτά που πετύχαμε. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ που κάνατε προσπάθεια να ολοκληρώσετε. Να περάσουμε στους επόμενους ε, συμμετέχοντες από την παρουσίαση. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της ε, Παγκόσμιας Τράπεζα, την κυρία Ματέρνοβα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε εξότιμοι βουλευτές. To be here and uh, for the World Bank to be involved. όπως είπε και η κυρία ε, Σουλτάνογλου, ξεκίνησε από το πιλωτικό πρόγραμμα για, κατά το αποκλεισμό των Ρωμά ε, μέσα στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ για την περιφερειακή πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα. Στόχος είναι να αντλήσουμε τα διδάγματα αλλά να συλλέξουμε και τα δεδομένα που δεν είχαμε ποτέ για την κατάσταση των Ρωμά. Θα μιλήσουν άλλοι συναδελφοί για τα δεδομένα. Εγώ θα σας μιλήσω πιο πολύ για τα διδάγματα τα οποία θεωρώ ότι έχουμε αντλήσει. Πρώτον, και η πιλωτική έρευνα και η έρευνα νοικοκυριών ε, δείχνει πόσο σημαντικά είναι τα δεδομένα, ιδίως έναν τομέα σε μια κοινότητα, για μια κοινότητα που ήταν τρομακτική έλλειψη δεδομένων. Και ιδίω εν καιρό κρίση βλέπουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δεδομένα και μα δίνουν τη δυνατότητα να δούμε αυτόν τον ε, πολύ ε, ύπουλο ε, συνδυασμό αυτής της κατάστασης, της στόχιας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον, σοκαριστικά στοιχεία έρθαν στο φως ο Γιάννης θα μας τα πει, ε, είναι από τον Οργανισμό Θεμελιωτών Δικαιωμάτων. Θα έχετε βέβαια όλη την έκθεση και τα στοιχεία. Μια πρόγευση θα την λάβετε σε λίγα λεπτά πάντως. η έρευνα νοικοκυριών και η πιλωτική έρευνα του Κοινοβουλίου μας έδωσε ήδη πολύ σημαντικά διδάγματα, πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση, συνάδελφος από την Παγκόσμια Τράπεζα θα σας τα πει, αλλά και στην ανακοίνωση που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα έχετε και εκεί κάποια στοιχεία. Κάτι που θα ήθελα εγώ να αναφέρω έχει να κάνει με το εξή. Μία από τις συνιστώσεις του πιλωτικού προγράμματος είχε να κάνει με τις μικροπιστώσεις ως έναν τρόπο που θα δώσει δυνατότητα στους Ρωμά να χρηματοδοτήσουν την αυτοαπασχόληση σε καιρούς μεγάλης ανεργίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που είδαμε με όλη αυτή την κρίση είναι ότι οι μικροπιστώσεις ουσιαστικά έχουν να κάνουν μόνο με ένα υποσύνολο, με ένα μικρό κομμάτι της κοινότητας των Ρωμά. Αλλά οι ανάγκε του είναι πάρα πολύ σημαντικέ για αυτό τον, την οικονομική ένταξη, όπω την αποκαλούμε, financial inclusion. Υπάρχουν ε, πολύ περιθωριοποιημένοι Ρωμά και η κατάστασή του προσωμιάζει χώρες ε, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, ε, στα βάθη του αναπτυσσόμενου κόσμου, σαν να μην είναι στην ε, σαν να μην είναι στο κέντρο της Ευρώπης αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Πέραν τώρα των δεδομένων, είναι ενδιαφέρον να έχουμε στατιστικά στοιχεία, να δούμε πώς ζουν οι Ρωμά, αλλά κάτι άλλο το οποίο βρήκαμε και είναι σημαντικό, είναι ότι με αυτά τα εργαλεία μπορούμε να χαράξουμε τις πολιτικές μας. Σε ό,τι αφορά την κοινότητα των Ρωμά, είναι γεγονός ότι πολλές πολιτικές προέρχονται μόνο και μόνο από κάποιες ε, απόψεις, πιστεύω, πεπιθήσεις, ε, ίσως και προκαταλήψεις και όχι από την πραγματικότητα, δεν βασίζονται στην πραγματικότητα. Γι' αυτό χρειάζονται στοιχεία. Είναι μια μυστηριώδης κοινότητα που κανείς ε, δεν την κατανοεί απόλυτα, άρα εάν κάποιος ε, κάνει μια κατάτμιση ε, των πολιτικών, παιδεία, στέγαση κτλ. και δει ε, όλα αυτά σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχουμε, τότε μπορεί να χαράξει τις βέλτιστες πολιτικές. Και αυτό ήταν ένα όφελος από αυτό το εγχείρημα που ξεκινήσαμε. Όπως ανακοίνωσε και, στη, η Κομισιόν, επιθυμεί και δίνει και εντολή στον Οργανισμό Θεμελιών Δικαιωμάτων να υλοποιήσει τις στρατηγικές ένταξης στον Ρωμά. Και αυτό είναι και ένα τομέα που πιστεύω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Να καλέσει δηλαδή τα κράτη-μέλη, είτε αυτή την πεποίθηση ότι απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, εθνικώ απομαδοποιημένε στατιστικές, να το υπερπηδήσει αυτό το εμπόθιο και να συλλέξει πλέον τέτοια στατιστικά στοιχεία ώστε να μπορεί η πολιτική να ε, χαράσεται βάση στοιχείων συγκεκριμένων και ή δυνατόν να προβεί σε κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές ενέργειες. Παραδείγματος χάρη ένα λεγόμενο booster sample, να έχουμε μια δηματοληψία που θα την προσθέσουμε στην ε, έρευνα για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης ε, την έρευνα ΣΥΛΚΑ που διεξάγεται σε αιτήσια βάση από τα κράτη-μέλη και τα στοιχεία τα σχετικά υποβάλλονται στη Eurostat που τα χρησιμοποιεί μετά για την χάρεψη τη χάραξη της πολιτικής. Να δούμε πού ζουν οι φτωχές κοινότητες, παραδείγματος χάρη. Και έχουμε και μια πρωτοβουλία της ΓΔ περιφερειακής πολιτικής που έδωσε εντολή στην Παγκόσμια Τράπεζα να χαράξει αυτούς τους λεγόμενους χάρτες φτώχειας, όπως τους ε, ονομάζουμε. Έτσι λοιπόν θα εκπονήσουμε αυτούς τους χάρτες τα επόμενα χρόνια που θα αποτελέσουν και μία βάση για να εντοπίσουμε που ζουν οι πιο φτωχοί συμπολίτες μας. Και κάτι τελευταίο. Μια σαρπαστική στιγμή για θέματα που έχουμε κάνει με την ένταξη των Ρώμα. Έχουμε την ιστορική ευκαιρία αυτή τη στιγμή στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων πραγματικά να κάνουμε τομή ε, στην ε, ένταξη των Ρωμά. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα υπάρχει πολιτική ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση και εδώ ε, και στα άλλα θεσμικά όργανα, αλλά και στις εθνικές κυβερνήσεις για την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ένταξη των Ρωμά. Έχουμε στοιχεία, οι χώρες θα έχουν επίσης πόρους στη διάθεσή τους, θα εισρέψουν πόροι, θα εισρέψουν κονδύλια και από χθε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ε, στις συστάσεις αναχώρα η ένταξη των Ρωμά συνδέεται στις δυνατότητες ε, των χωρών που έχουν μεγάλους πληθυσμούς Ρωμά για να επιτύχουν τους στόχους του 2020. Δηλαδή μπαίνει στο ανώτατο επίπεδο, ψηλά ε, στις προτεραιότητες της Ατζέντα 2020. Τελευταία πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Εσείς ε, θα εγκρίνετε τους κανόνες με τα διευθυντικά ταμεία όπου να είναι. Η ένταξη των Ρωμά στο Συμβούλιο ήταν περιορισμένη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέχρι τώρα. Είναι νομίζω στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διευρύνεται το πεδίο εφαρμογή και σε ό,τι αφορά την ε, ε, εξάντε αιρεσιμότητα για την κοινωνική ένταξη και τον αποκλεισμό, είναι στα χέρια σα η ένταξη των αρμών να μπει σε όλα τα ταμεία και όχι μόνο στο κοινωνικό. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ και τώρα να περάσουμε στο τρίτο τμήμα της παρουσίασης σε ό,τι αφορά της δυνατότητας ε, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο κύριο Δημητρακόπουλος. Πέντε λεπτά έχετε στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι το συντομότερο δυνατό όσο το πιο γίνεται πιο σύντομος, να σας πω ότι έχει γίνει. Η Task Force ε, δημιουργήθηκε το 2010 το Σεπτέμβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση και βρήκε ότι υπήρχαν προβλήματα σε αρκετούς τομείς και σε ό,τι αφορά τη διαθέσιμότητα ε, στοιχείων αδιάσυστων για τους Ρωμά. Η πρόκληση που αντιμετωπίσαμε ήταν ότι το θέμα της ε, ένταξης των Ρωμά είναι ένα πολυδιάστατο θέμα, το οποίο, όπως είπατε κι εσείς, ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενοποιημένη προσέγγιση για θέματα και φτώχειας, αλλά και ανθρωπινών δικαιωμάτων. Να μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία των πολιτών έχει σε πολλές περιπτώσεις τονίσει ότι η έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη, η έλλειψη δικαιοσύνης, ισότητας οδηγούν σε ένδια, περιθωριοποίηση και τελικά ε, καταλήγουμε στην σημερινή κατάσταση των Ρώμα. Η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ανέπτυξε ένα οκταετές πρόγραμμα το οποίο θα συμπεριλάβει δύο κύματα της έρευνας τα οποία έγιναν ε, στην ε, διάμεση θεώρηση για την στρατηγική του 2020 για να μετρηθεί η πρόοδος. Αυτό δεν επαρκεί και τα κρατημέλη θα ε, υποστηριχθούν και το έχουμε ξεκινήσει αυτό για να αναπτύξουν τα εργαλεία παρακολούθησης για την ε, παραγωγή συγκριτικών στοιχείων για να δούμε ποια κράτη-μέλη τα πηγαίνουν καλύτερα και πού μπορούν να βελτιωθούν τα κατάσταση. Παράλληλα θα πρέπει να κατανοήσουμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Άρα από το 2013 μέχρι το 2016 θα κάνουμε ε, ποιοτική εργασία όσο πιο κοντά γίνεται στον πολίτη και στις τοπικές αρχές για να δούμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Πολλά έχουμε ακούσει για τον τρόμα. είναι εθνική μειονότητα, κατά πόσο είναι δυνατόν να συλλέξουμε εθνοτικά στοιχεία. Φυσικά υπάρχει ιστορική εμπειρία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη, αλλά αφετέρου υπάρχει και ανάγκη να υπάρξουν τέτοια ενοποιημένα δεδομένα για να υπάρχουν ε, αποτελεσματικές πολιτικές. Η προστασία των δεδομένων είναι θεμελιώδες δικαιωμάτων. Αλλά σήμερα έχουμε τις σχετικές διατάξεις, τις σχετικές δομές, προκειμένου να προστατεύσουμε αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα και να συλλέξουμε σημαντικά στοιχεία. Έχουμε συνοπτικές, συνοπτική ε, νομοθεσία και έχουμε και τις αρχές προστασίας των δεδομένων. Για να σας πω τι γίνεται στην έρευνα. Ότι και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και σε χώρες όπως την Ιταλία, την Πορτογαλία ε, υπάρχει αυτή η συνεργασία. Καλύπτει μεγάλον αριθμό Ρώμα και μη Ρώμα και μας επιτρέπει να δούμε ποιε είναι οι διαφορές και ποιε είναι οι δημορφίε των κοινοτήτων αυτών. Έχουμε εκπροσώπους των τοπικών αρχών ε, στα μέρη που έλαβε μέρος ε, χώρα η έρευνα και θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα ε, μέσα στο έτος. 11 κράτη-μέλη συμμετείχαν, αλλά η UNDP συμμετείχε και σε τρίτες χώρες στην, στα Βετικά Βαλκάνια, και στη Μολδαβία. Να σας δείξω κάποια παραδείγματα τώρα για το πόσο ε, εκτενής ήταν η εθνική δειγματοληψία. Δεν πήγαμε μόνο σε τομείς ε, με μικρούς οικισμούς, όχι. Στις διάφορες χώρες ε, πήγαμε στις πράσινες κουκίδες όπου βλέπετε στη διαφάνεια σε κοινότητες Ρωμά και αυτό δείχνει πόσο ατεκμηριωμένη είναι η έρευνα στη Γαλλία. Ε, πήγαμε σε κοινότητες όπου ζουν συνήθως οι Ρωμά και τα αποτελέσματα καταρχάς θα εστιάζονται στην κατανομή αναηλικία. Αυτό θα πρέπει φυσικά πιο λεπτομερώς να, να εξεταστεί, αλλά δείχνει ότι είναι υψηλά τα ποσοστά γονιμότητας και θνησιμότητας σε σχέση με τους Ρωμά. Ε, κόκκινη είναι η Ρωμά, μπλε η μη Ρωμά στην διαφάνεια. Να σας ε, παρουσιάσω αν και ο συνάδελφος θα σας δείξει πιο πολλές πληροφορίες, να σας δείξω ε, με κόκκινο την ε, χώρα μου, την Ελλάδα, που έχει τον χαμηλό ποσοστό ε, για την ηλικία 4 έως 6 έτη συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση. Βλέπετε λοιπόν ότι μας ανησυχεί ιδιαίτερα ο αριθμός παιδιών που βρίσκονται σε ηλικία υποχρεωτικής παρακολούθησης ε, του σχολείου που δεν παρακολουθούν όμως το σχολείο. Είναι σε κάποιες περιπτώσεις πάρα πολύ υψηλό ποσοστό και πάλι στην Ελλάδα άνω του 30% είναι το ποσοστό αυτό. Αυτό που μας ανησυχεί και στο πλαίσιο της κρίσης είναι οι ενήλικες 20-24 ετών που παρακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση. Βλέπετε ότι το ποσοστό των Ρωμά που δεν έχουν την ικανότητα να ανταγωνιστούν στην αγορά εργασίας είναι πολύ υψηλό. Τέλος, ε, να δούμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά τη κριτική μεταχείριση. Βλέπετε το 2008 που έγινε η μελέτη, η ανάλυση καταδεικνύει ότι τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Είναι υψηλά τα ποσοστά διακριτικής μεταχείρισης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πολλοί από τους ερωτηθέντες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν ήξεραν καν ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία για την διακριτική μεταχείριση. Τέλος, θα ήθελα σε μια διαφάνεια να σας δείξω κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Όταν ρωτήσαμε τους επίσημους εκπροσώπους των τοπικών αρχών αν γνωρίζουν ότι υπάρχει ε, νομοθεσία που προστατεύει κατά της διακριτικής ε, μεταχείρισης βάσει εθνοτικής προέλευσης, από ό,τι βλέπετε σημαντικός αριθμό σε όλα τα κράτη-μέλη δεν ήξερε καν ότι υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Άρα, συνολικά, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πλέον επαρκή στοιχεία που μας οδηγούν στην... Ε, τα μέτρα για τη συμπερίληψη των Ρωμά πλέον. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το δεύτερο τμήμα της ε, παρουσίασης από την Παγκόσμια Τράπεζα. Ο κύριος Τελάτινο ο υπεύθυνο, ο οποίος και θα μας κάνει μια παρουσίαση ε, εξ ονόματος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σας παρακαλώ πολύ, όχι παραπάνω από 5 λεπτά. Thank you. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, εξότιμα μέλη, που με επιτρέπετε να παρουσιάσω, να σας παρουσιάσω κάποιες ε, συστάσεις για πολιτική που από την επισκόπηση αυτή, από την έρευνα. Θα είμαι πολύ σύντομος. Υπάρχουν τέσσερα βασικά μηνύματα που θα ήθελα να σας παρουσιάσω σήμερα. Το πρώτο είναι ότι η αρχική εκπαίδευση και η μέρημνα των παιδιών είναι βασικό στοιχείο για να σπάσει αυτός ο κύκλος ε, της φτώχειας. Υπάρχουν στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο και όπως σας δείξω και σε ένα λεπτό υπάρχουν και σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την έρευνα για τους Ρωμά ότι αυτό ισχύει και στην κάλυψη της, του χάσματος γενεών και για τους Ρωμά. Βλέποντας την έρευνα βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστιο κενό στα αποτελέσματα για την αρχική εκπαίδευση και τη μέρη των παιδιών και στον υπηαγωγείο και στο σπίτι. Και δείχνει τέλος η έρευνα διάφορες επιλογές πολιτικής που μπορούν να εφαρμοστούν για να αντιμετωπιστεί το κενό. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται ευαισθητοποίηση των, γονέων, να καλυφθεί το κενό στην, της γνώσης θα πρέπει να αφαιρεθούν ε, οι φραγμοί όσον αφορά το κόστος και θα πρέπει να δίνονται επιδοτήσεις για να υποστηρίζονται οι γονεί για να πηγαίνουν τα παιδιά στον υπηαγωγείο και να υποστηρίξουν μετά τους γονείς στο σπίτι ε, ούτως ώστε να δώσουν κάποια κίνητρα ε, ενδιαφέρον στα παιδιά τους να μάθουν. Θα σας δώσω κάποιες διαφάνειες. Αυτή είναι μια διαφάνεια από μια έρευνα που έκανε το Lancet για την αρχική εκπαίδευση των παιδιών. Εάν δεν καλυφθούν ανισότητες και κενά, όσον αφορά την κακή διατροφή, πριν τη γέννηση των παιδιών, μέχρι τα πρώτα χρόνια των παιδιών, θα παραμείνει ένα κενό που θα εξακολουθεί να εφίσταται κατά τη διάρκεια της ζωής του παιδιού. Με άλλα λόγια, πρέπει να επενδύσει κανείς νωρίς, διότι θα έχει μεγάλη απόδοση μελλοντικά. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ φτωχών και πλούσιων όσον αφορά την πρόσβαση στην συγκρίνεται τους Ρωμά με τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι πολύ μεγαλύτερη διαφορά των Ρώμα με τους άλλους από ό,τι διαφορά μεταξύ πλουσίων και φτωχών στον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά τα αποτελέσματα, όσον αφορά τις γνώσεις των μικρών παιδιών. Βασικό μήνυμα από την έρευνα του Lancet. Χρειάζεται έγκαιρη επένδυση, διότι η επένδυση σας δίνει κέρδη μακροπρόθεσμα για την ένταξη. Αυτό είναι το ιστορικό. Δίνονται και λεπτομερείς πληροφορίες. Ερώτημα βασικό. Ίσως οι Ρωμά δεν θέλουν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους. Μήπως αυτό συμβαίνει. Αυτό δεν απορρέει από την ερεύνα. οι προτιμήσεις την εκπαίδευση των παιδιών τους μοιάζουν με τις προτιμήσεις ε, των, ε, της πλειοψηφίας των πληθυσμών στις περισσότερες χώρες που μένουν. Η κρίση. Την έχουν όλοι υπόψη. Τη βλέπουμε και στην έρευνα. Ο συνάδελφος Αντρέη από το UNDP θα αναφερθεί λεπτομερέστερα σε αυτό. Ποσοστά σωστά ε, οικογενειών που πεινούν κάθε μήνα. Από 23% μέχρι 60% ποικίλει το ποσοστό. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο όσον αφορά την κακή διατροφή των παιδιών. Πάνω από 50% των παιδιών στη Βουλγαρία, Ρουμανία και τη Σλοβακία δεν έχουν ένα βιβλίο ή έχουν ένα βιβλίο στο σπίτι. Τα παιδιά που πήγαν στον υπηαγωγείο και σε ενήλικους και νέους στις ίδιες κοινότητες με παρόμοιο ιστορικό και συγκρίνουμε αυτούς που πήγαν νηπιαγωγείο με αυτούς που δεν πήγαν, βλέπουμε στη Τσεχική Δημοκρατία, στη Σλοβακία, όπου πολλά μικρά παιδιά πάνε σε ειδικά σχολεία για άτομα με αναπηρίες. Βλέπουμε ότι το νηπιαγωγείο καλύπτει τα κενά από μισό μέχρι ένα τρίτο. Στα παιδιά που έχουν πάει στο νηπιαγωγείο είναι πολύ πιο σίγουρο ότι θα καλύψουν, θα ολοκληρώσουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και τα καταφέρουν καλύτερα αργότερα στη ζωή τους. Έχουμε κακά και καλά μαντάτα όσον αφορά τα κενά. Τα άσχημα μαντάτα. Οι διαφορές στις περισσότερες χώρες είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όσον αυτή την πρόσβαση ε, στα νηπιαγωγεία, με εξαίρεση Ουγγαρία και Ισπανία. Αν δείτε την πολιτική της Ουγγαρίας, προσπαθεί να υποστηρίξει τους στοχούς γονείς. Να μην υπάρχει πρόβλημα κόστους και να δίνει επιδοτήσεις από το 2009 για να μπορούν τα παιδιά να πήγαν στην υπηαγωγία. Γιατί οι γονείς δεν βάζουν τα παιδιά τους στην υπηαγωγία. Απαντήσεις. Βασικός λόγος. Το παιδί είναι πολύ μικρό. Μπορούν να καλύψουν ανάγκη στα παιδιά. Και έχουν λόγους να μεγαλώσουν τα παιδιά στο σπίτι. Αυτό. Το κόστος. Άλλη απάντηση. Το πόσο δαπανηρό ποικίλει κατά χώρα. Πολλοί γονεί είπαν ότι θα επανεξέτασαν δυνατότητα να πάω στον υπηαγωγείο τα παιδιά αν ήταν δωρεάν και αν υπήρχαν και κάποιοι, αν διδασκόταν και ε, Ρωμά στα σχολεία. Τα παιδιά θέλουν να εκπαιδευτούν τα παιδιά. Οι γονεί θέλουν να εκπαιδευτούν τα παιδιά. Θέλουν τα παιδιά τους να έχουν την ίδια εκπαίδευση όπω ο υπόλοιπο πληθυσμό. Όμω προτιμούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στο σπίτι. Και ε, θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε το, τους γονείς ώστε να πιστέψουν τα παιδιά στην νηπιαγωγία, να τα βάλουν στην νηπιαγωγία. Θέλουμε να συμμετέχουν στη διαδικασία της εκπαίδευσης νηπιαγωγία οι γονείς και θέλουμε να μην υπάρχει πρόβλημα κόστους, να δίδονται επιδοτήσεις για να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο. Τέταρτον, θέλουμε να υποστηρίξουν τους γονείς που δίνουν εκπαίδευση στο σπίτι. Αυτά έχουν εφαρμοστεί σε κάποια μέρη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και νομίζω ότι και η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει. Ευχαριστώ κύριε Ντελάτ. Δεύτερο κομμάτι της παρουσιάσεως του UNDP, ο κύριος Ιβάνοφ. Παρακαλώ ένα πεντάλεπτο, ούτε λεπτό παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπόσχομαι να μην ξεπεράσω αυτά τα πέντε λεπτά. Let me start where we have this technical moment with uh, one να ξεκινήσω με μια γενική παρατήρηση. Όταν προπαρασκευάσαμε ε, την έκθεση με την ανάλυση των πρώτων δεδομένων, συζητούσαμε με τους υπεύθυνου από το Γραφείο Επικοινωνίας και με ρώτησε ένα συνάδελφος ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτή την έρευνα. Για να σας πω την αλήθεια, δεν θα έλεγα ότι το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Ρώμα είναι πιο φτωχή από τους άλλους. Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανεργία και μακροχρόνια ανεργία και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτό που εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε περισσότερο είναι ότι η διαφορά μεταξύ ε, επιτυχών ή μη επιτυχών δεν έχει να κάνει με τα νέα κράτη-μέλη, τα παλιά κράτη-μέλη ή με κράτη-μέλη και μη κράτη-μέλη. Και με αυτό θα ξεκινήσω, γιατί τα δεδομένα τα οποία έχουμε και που συνοψίζονται στην έκθεση, ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να δείχνουν την κορυφή του παγόβουνου. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα χρειαστεί και ελπίζω να συνεχιστεί μια διεξοδική ε, συνεχιζόμενη ανάλυση των στοιχείων. Και κυρίως αυτό που χρειάζεται είναι να διδαχθούμε από τα μηνύματα που μας δίνουν τα στοιχεία και να κάνουμε πράγματα στην πράξη. Διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Αυτό λένε τα στοιχεία. Ο στόχος όλου του εγχειρήματο είναι να αλλάξει κατάσταση και αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Κάτι το οποίο λοιπόν προκύπτει ξεκάθαρα είναι η ανεργία. Βλέπετε σε αυτό το γράφημα, παραδείγματος χάρη στην Ουγγαρία, αν δείτε πιο προσεκτικά τα στοιχεία, θα δείτε ότι πάνω από το 41% των ανέργων ε, ε, Ρωμά είναι ανέργοι για πάνω από από χρόνια. Όντας λοιπόν λοιπόν χρόνια εκτός ε, αγοράς εργασίας, τι δεξιότητες μπορεί να έχει κάποιος. Και είναι και μεγάλο ποσοστό που δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Νομίζω ότι αυτό δεν χρήζει καν σχολιασμού. Παγιδευμένη στην ανεργία είναι η Ρωμά και αυτό το βλέπουμε ε, και σε κράτη-μέλη της Ένωσης και σε χώρες εκτός Ένωσης. Ε, Παραδείγματο χάρη, ποιο είναι το μέλη αυτών που δεν έχουν εργαστεί ποτέ μεταξύ ε, του ενεργού πληθυσμού, του παραγωγικού δυναμικού ηλικία, δηλαδή από 15 έως 24. Βλέπετε τις τα γραφήματα, βλέπετε τις γραμμές αυτές, τις θαλασσιές. Βλέπετε λοιπόν και πάλι να προκύπτει το ερώτημα. Πώ μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν μετά μια θέση, δουλε... μια θέση εργασία. Εδώ βλέπουμε ακόμη ένα γράφημα, αλλά αφορά την Κροατία αυτή τη φορά. Αριστερά, το αριστερό τετραγωνίδιο. Βλέπουμε τους Ρωμά οι οποίοι έχουν μια θέση εργασίας. Και αριστερά, ε, δεξιά μάλλον, είναι η μη Ρωμά που είναι άνεργη. Επίσης βλέπουμε ότι και οι γυναίκες είναι περισσότερες σε σχέση με τους άντρες. Τώρα, διαφορές οδήματο. Σε όλες τις χώρες. Και οι δαπάνες και τα έσοδα είναι μικρότερα. Για τους Ρωμά και τους ε, γείτονες μη Ρωμά και το τονίζω γείτονες, γιατί αυτοί έχουν το ίδιο κοινωνικό οικονομικό περιβάλλον δηλαδή αν υπάρχει ύφεση, αν υπάρχουν ε, λίγες ευκαιρίες απασχόλησης και ούτω καθεξής. Άρα έχουν ε, και ένδια, στέρηση ε, βασικών αγαθών κτλ. Και αυτό βλέπουμε στο γράφημα αυτό. Αυτές οι μαύρες γραμμές είναι οι μέση όροι. Αν συγκρίνουμε τους εθνικούς μέσους όρους με την κατάσταση των Ρωμά, βλέπουμε ότι σε περισσότερες περιπτώσεις έχουμε διπλάσια ή τριπλάσια ε, στέρηση για τους Ρωμά. Επίσης, η πείνα που αναφέρθηκε είναι πράγματι ένα πρόβλημα, είναι ένα ζήτημα και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ βλέπετε το παράδειγμα της Ρουμανίας, αλλά νομίζω ότι σε όλες τις χώρες τα πράγματα είναι παρόμοια. Το 61% των Ρωμά της Ρουμανίας έχουν πει ότι πάνε νηστικοί στο σπίτι το βράδυ να κοιμηθούν γιατί δεν μπόρεσαν να αγοράσουν τρόφιμα. Ποσοστά φτώχειας. Η Ρώμα δεν είναι απλά φτωχότερη, αλλά είναι και πιο βαθιά βυθισμένη στη φτώχεια. Τελευταίο σλάιτ είναι οι μεταναστευτικέ στρατηγικές. Οι Ρωμά που βλέπουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ποιες είναι οι τρεις χώρες προορισμού εδώ για τους Ρωμά τη Σλοβακία είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τσεχία και η Γερμανία. Δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα σλάιτ ε, χρήζουν περαιτέρω αναλύσεων ή ερμηνείας. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει πλέον είναι να ξεπεράσουμε κάπως ε, και αυτά τα γραφήματα και ε, τις διαφάνειες. Ξέρουμε τους παράγοντες που προκαλούν την κατάσταση, ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση, τι πρέπει να κάνουμε, τη δουλειά μας. Πολύ απλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει και αυτή μια δήλωση και μετά θα έχουμε ε, τη συζήτηση. Νομίζω ότι Έχουμε εδώ την εκπρόσωπο, ε, το Διευθυντή για την Ισότητα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της ΛΥΜΠΕ, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Ε, είμαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω εν συντομία το εξής. Καταρχάς να πω ότι είμαι ευγνώμων προς το UNDP, προς την ε, Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και για την Παγκόσμια Τράπεζα για την, για την ε, προσπάθεια που έχουν καταβάλει σε ό,τι αφορά την ε, έρευνα αυτή και μας ε, δίνουν τεκμηριωμένα στοιχεία τα οποία μας χρειάζονται. Υποστηρι... Επίσης ευχαριστούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υποστήριξε το πολιτικό project επί του οποίου βασίστηκε και φυσικά είμαστε ευγνώμονες και στους συναδέλφους μας, από την ε, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής γιατί έχουν διαχειριστεί το σχετικό πολιτικό project σε συνεργασία με τις ε, τρεις αυτούς φορείς που ανέφερα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα στοιχεία αυτά σε ό,τι αφορά την ε, παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας ε, των πολιτικών για τους Ρωμά και χαιρόμαστε που διαπιστώνουμε ότι η έρευνα αυτή πλέον διατίθεται ένα έτος μετά από την έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προετοιμαστεί. Θα είναι πραγματικά καθοριστική τα επόμενα χρόνια για μας τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν σε ό,τι αφορά και το διάλογο με τα κράτη-μέλη. Θα μιλήσουμε και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλώς με τα κράτη-μέλη, αλλά και με τα εθνικά σημεία επαφής και τα σχετικά δίκτυα που σκοπεύουμε να συστήσουμε όπως αναφέραμε και στην ανακοίνωση την οποία εγκρίναμε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου έγινε η αξιολόγηση των πολιτικών ε, ένταξη των Ρώμα, την οποία μας διαβίβασαν τα κράτη-μέλη, σκοπεύουμε να εξετάσουμε στενά τους τέσσερις τομείς πολιτικής, όπως και τον τομέα της ε, μη διακριτικής μεταχείρισης ε, και αυτά θα γίνουν βάση των τεκμηριωμένων στοιχείων της έρευνας. Αφετέρου δεν μπορούμε παρά να αισθανόμαστε σοκαρισμένοι με την πραγματικότητα που αποτυπώνει αυτή η έρευνα. Είναι μια ανησυχητική εικόνα. Μια ανησυχητική εικόνα τάσεων που επιδεινώνονται σε πολλά κράτη-μέλη. Και χρειαζόμαστε κατεπίγουσα και συγκεκριμένη δράση. Αυτό θα βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη τον επόμενο καιρό. Και θα πρέπει απαραίτητος να υπάρξουν αποτελεσματικές δράσεις για σημαντικά αποτελέσματα την επόμενη περίοδο. Και πάλι λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις φορείς ε, και υπομονούμε και προσβλέπουμε σε μια ε, ενδεχόμενη παρουσίαση και συζήτηση της ανακοίνωσης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενδεχόμενες στρατηγικές από τα κράτη-μέλη, όπου θα κοιτάξουμε πιο ενδελεχώς κάποια επιμέρους στοιχεία, μια συζήτηση την οποία θα διοργανώσει το Κοινοβούλιο. Μάλιστα, πολύ σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκέντς έχει τώρα το λόγο για να κάνουμε την συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφενός, χαίρομαι ιδιαίτερως που γίνεται η συζήτηση αυτή και έγιναν αυτές οι παρουσιάσεις γιατί εδώ και καιρό αναμένουμε σχετικά στοιχεία και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι χωρίς τα τεκμηριωμένα στοιχεία δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε το τι πραγματικά συμβαίνει επί τόπου. Είναι μεγάλο επιτεύγμα το ότι υπάρχουν πλέον στρατηγικές, εθνικές στρατηγικές και το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν εύκολο, αλλά πλέον βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο εκκίνησης. Μεγάλο ερώτημα. Το μεγάλο μου ερώτημα είναι το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Σε συνέχεια της έρευνας αυτής θα γίνουν και άλλες δύο έρευνες σε κάποια χρόνια, αλλά νομίζω ότι πολύ σημαντικό θα είναι αφενός να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή των πολιτικών και το μοναδικό ερώτημα που ανέκυψε όταν διάβαζα τις στρατηγικές είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις μου φαίνεται κατάλογος ε, ευσεβών πόθων. Σε, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρχε συγκεκριμένο συγκεκριμένη χρηματοδοτική πόρη που συνδέονται με τις επιθυμίες αυτές. Άρα το θέμα είναι πόσο θα μπορέσει να παρακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τι συμβαίνει επί τόπου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι πραγματικότητες που θα διαμορφωθούν κατά αναλογία με τις στρατηγικές. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι τεράστιες οι διαφορές. Ε. Οι στρατηγικές αποτυπώνουν μια πολύ καλύτερη εικόνα από τη είναι στην πραγματικότητα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πιο πολλά πράγματα σχετικά με το τι σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον και τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση των ε, πολιτικών αυτών. Κάτι άλλο, ένα άλλο ερώτημα. Οι πόροι αυτοί και τα μελλοντικά λειτουργικά προγράμματα καλύπτονται από τα προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο λοιπόν για να ελέγξει την αιρεσιμότητα εξάντε Νομίζω λοιπόν ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι καθοριστικός. Δεν χρειάζεται να συνεχίσω. Νομίζω ότι είναι και περιορισμένο το χρονικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Γιάροκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους ε, τους φορείς που μας παρουσίασαν τα στοιχεία αυτά, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε προκαταρκτικό στάδιο, υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία. Τα βασικά στοιχεία που ήθελα να αναφέρω είναι τα εξή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι καλύπτονται οι χώρες της έκτης διεύρυνσης και βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να ε, ανταποκρίνονται σωστά αυτές οι χώρες στις σχετικές ε, ανάγκες. Οι θεματικές εκθέσεις θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως αναφέρετε στην εκθέσή σας, για τους τέσσερις θεματικούς τομείς τους οποίους ε, υπογραμμίσαμε, θα πρέπει να κινηθούμε σε βάθος για να αναβαθμίσουμε τα πορίσματα, να αναβαθμίσουμε και τα project. There is also Επίσης, υπάρχει άλλος ένα σημαντικό τομέα, τον οποίο προτείνεται να γίνει ερευνά. Τα κεφάλαια μεθοδολογίας και εισαγωγή μιλούν για την υποδομή και την γειτονία, αλλά σχετικά πορίσματα δεν τα βρήκα στην έκθεση. Μιλήστε μας λοιπόν για τα αποτελέσματα αυτά. Επίσης πείτε μας ε, πόσοι η μεθοδολογία συνδέεται με τους εταίρους του τέταρτου ομίλου και ποιοι είναι οι επόπτες του κεφαλαίου αυτού. Αναφερθήκατε στη σημασία του χάρτη ένδυας, του χάρτη κρίσης, ε, όπως αναφέρατε τότε. Θα θέλαμε ένα τέτοιο χάρτης να υπάρχει για όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν έγινε, αλλά ελπίζουμε ότι τα... θα γίνει έρευνα και στα υπόλοιπα 16 κρατημέλη. Λόγω των περιορισμών που έχουμε, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω εκ νέου ότι η ιδέα για το χάρτη κρίσης και ένδυας που είχαμε αρχικά και που αναφέρεται στις εκθέσεις του Κοινοβουλίου προαπαιτεί έρευνα με όλους τους κοινωνικονομικούς φορείς. Άρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα, την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, περιβαλλοντικών υπηρεσιών, υποδομές μεταφορών. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία λείπουν από την έρευνα. Έγινε πολύ, έχουν γίνει πάρα πολλή έρευνα για τους Ρώμα τα τελευταία 20 χρόνια και σήμερα ήταν η πρώτη εμπειρία που είχα πραγματικά σε ό,τι αφορά θέματα διακριτικής μεταχείρισης. Αναφέρατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για τους Ρωμά σε ό,τι αφορά τη διακριτική μεταχείριση βάσει εθνοτικής προέλευσης. Αυτά τα επανέλαβε και η κυρία Ρέντινγκ. But that, it was very important on the... Πέρα από αυτά, ήταν πάρα πολύ σημαντικό στη διαφάνεια της Παγκόσμιας Τράπεζας το ότι είδαμε ποια είναι η κατάσταση για τα παιδιά των Ρώμα και ότι οι δέκα βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν ε, την κατάστασή τους δεν ε, περιλαμβάνουν και την διακριτική μεταχείριση. Κοιτώντα τα πραγματικά στοιχεία, είναι ενδιαφέρον το ότι βλέπουμε ότι αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα τα τελευταία 20 χρόνια, βάσει των οποίων καταστρώναμε και τις πολιτικές μας, πλέον διαψεύδονται. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε και για τα υπόλοιπα ερωτήματα να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα και για τους κοινωνικονομικούς παράγοντες που συζητήσαμε στην έκθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά σας και προσβλέπουμε σε μελλοντική συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστούμε κυρία Γιάροκα. Έχουμε άλλους τρεις ομιλητές στον κατάλογο που θέλουν να μιλήσουν. Σημαντικό να περιοριστείτε χρονικά, διότι ψηφίζουμε στις 12 και εξακολουθούμε να έχουμε και μεικτή συζήτηση, κοινή συζήτηση στο πιο ευαίσθητο θέμα πριν την ψηφοφορία. Ε, έχετε το υπόψη. Βοηθήστε μας. Ναι. Η κυρία Ντάνοκα. Θα είμαι συντομότατη. Uh, resolution on Roma, uh, I was also a reporter for strategy of European Union for non Για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη διάκριση και το θέμα των Ρώμα. Και έχουν προβλέψει θετικές δράσεις. Θετική διάκριση αποκαλείται στη ΣΥΠΑ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει στρατηγική για την αντιμετώπιση ενέργεια των Ρωμά. Στις συστάσει πρέπει να συμπεριλάβουμε την ανάγκη για έρευνα. Να δούμε πώς τα κράτη-μέλη και οι αρχές τους χρησιμοποιούν την προσέγγιση που αναφέρατε εδώ για να βελτιώσουν την κατάσταση. Το γιατί δεν πήγαν τα παιδιά στο σχολείο. Εξετάσατε τις γλωσσικές γνώσεις. Αν είναι εμπόδιο γνώσεις γλωσσών για τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Και κάτι άλλο σχετικό. Θα ήταν ενδιαφέρον να ξέρουμε Ποιε είναι οι μεταναστευτικέ ροέ εντό Ευρωπαϊκή Ενώση για τι οικογένειε στο Ρώμα. Πόσε οικογένειε δεν μένουν στη χώρα τη οποία την ηθαγένεια κατέχουν. Αυτό ήταν ενδιαφέρον να το γνωρίζουμε. Ο κύριος Μπρόγκς. Ευχαριστώ. Η Ρώμα φαίνεται να γίνεται της μόδας και να μην είναι της μόδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ρώμα τελικά σε ομιλίες και σε έγγραφα αναφέρονται σαν να μην άτομα. Αναφέρονται παθητικά, σαν να είναι άτομα στα οποία τους κάνουν πράγματα αυτό, όχι αποκλεισμό, στέρηση. Ή ότι πρέπει να τους κάνουμε κάποια πράγματα, να τους δίνουμε χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ποτέ δεν αναγνωρίζουμε ότι κάνουν πράγματα για αυτούς ή σε αυτούς σαν να μην θεωρούμε ότι έχουν την ικανότητα. Πόσοι ευρωβουλευτέ συναντούν, ε, έχουν συναντήσει Ρώμα. Ίσως να βλέπω κάποια φωτογραφία σε κουτί με σοκολατάκια. Εγώ έχω συναντήσει Ρώμα. Ξέρω και τα καλά δύο από αυτού και τα κατάφερα μια χαρά. Δείχνει ότι καμιά φορά οι Ρώμα μπορούν να δράσουν επωφελώς για τους αυτούς τους. Καμιά φορά κάνουν πράγματα σε αυτούς τους και ο ένας τον άλλον που πόρα απέχουν από ευεργετικά αποτελέσματα. Πριν δύο χρόνια κάναμε ακρόαση αυτή την ε, επιτροπή για το εμπόριο λευκής αρκός ε, άνδρες, ε, για, συγγνώμη, γυναίκες και παιδιά. Κάποια πληθυσμιακή ομάδα είχε εκπροσωπηθεί δυσανάλογα μεταξύ εκείνων που ασκούσαν το εμπόριο και εκείνων που ήταν θύμα του εμπορίου. Η απάντηση αφής από τη Europol στο ερώτημα. Η απάντηση ήταν η Ρωμά. Οι άντρε Ρωμά εμπορευόταν γυναίκες και κορίτσια Ρωμά για πορνεία. Αν το αφισβητείτε αυτό, τα πάτε στο Στασβούργο, κοιτάξτε ανατολικά στα, στους καταβλισμούς των Ρωμά και πιο κάτω θα δείτε κορίτσια Ρωμά και το χρησιμοποιώ σωστά κορίτσια Ρώμα που κάθονται δίπλα στο δρόμο και περιμένουν. Και οι αρχές του Στρασβούργου δεν έχουν κάνει τίποτα γι' αυτό και αυτό είναι τραγικό. Αναφέρθηκε πριν ότι έμοιαζε η ζωή τους με ζωή ανθρώπου στον κόσμο παρά κόσμου στην Ευρώπη. Ίσως διότι προέρχονται αρχικά, κατάγονται από τον τρίτο κόσμο. Όταν φέρνεις κόσμο από τον τρίτο κόσμο, αλλάζει τον κόσμο ή αλλάζει την Ευρώπη. Αυτό είναι το τρίτο ερώτημα που έχω από αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερζάτ. Εγώ δεν ε, βλέπω τους Ρωμά μόνο σε κουτιά από σοκολατάκια και ούτε μόνο δύο ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν έρχονται από τον τρίτο κόσμο. Παρ' όλα αυτά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές ε, για την πολύ ποιοτική τους δουλειά. Πράγματι, είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια μεγάλη εμβέλεια έρευνα για την κατάσταση των Ρωμά στην Ευρώπη σε έναν συγκεκριμένο αριθμό χωρών αρκετά διαφορετικών μεταξύ τους και αυτό το θεωρώ εξαιρετικό. Αυτό επιβεβαιώνει, όπως υπόθηκε άλλωστε, όλα τα στοιχεία τα οποία εμείς γνωρίζουμε ιδιαίτερα καλά στην Επιτροπή μας αυτή και στο Κοινοβούλιο κάτ' επέκταση. Οι χειρότεροι φόβοι μας, θα έλεγα, επιβεβαιώθηκαν. Και πράγματι αυτό θα αποτελέσει ένα εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό στα χέρια μας για το έργο που έχουμε να επιτελέσουμε σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών. Θα σας δώσω το παράδειγμα της χώρας που γνωρίζω καλύτερα, της Γαλλίας δηλαδή. Η εθνική στρατηγική που παρουσιάστηκε από τη Γαλλία υπολείπεται των πάντων και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Είναι κάτω από οποιαδήποτε προσδοκία. Είναι, τι να πω, ε, μία φενάκι όλα αυτά. Είναι σαν αυτοί που ταξιδεύουν να είναι ε, Γάλλοι και οι Ρωμά να είναι άνθρωποι που έρχονται από άλλα κράτη-μέλη. Ε, θα ήθελα να δω και τα στοιχεία, τα πιο αναλυτικά για την έρευνα στη Γαλλία, που έχει να κάνει με αυτό που εμείς λέμε, έτσι ονομάζουμε, Ρώμα, αλλά τον οποίο η κατάσταση είναι πολύ πιο δραματική από αυτή που φαντάζομαι ότι εσείς διαπιστώσατε. Σε σχέση με αυτούς που εμείς ε, ονομάζουμε «Jean de ανθρώπους που ταξιδεύουν, νομάδες, ε, περιπλανόμενους. Πώς θα συνεργαστούμε στο μέλλον, ώστε οι πολιτικές αυτές οι οποίες ε, βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης δεν θα παραμείνουν στα λόγια και θα αποτελέσουν τα θεμέλια συγκεκριμένων δράσεων. Και κάτι τελευταίο. Μεταξύ όσων άκουσα, αυτό το οποίο με εντυπωσίασε ιδιαίτερα και θα ήθελα να ακούσω περισσότερα, ήταν το γεγονός ότι οι διαφορές τις οποίες διαπιστώσατε δεν είναι διαφορές μεταξύ των νέων κρατών μελών και των παλαιών ε, κρατών μελών ή μεταξύ ε, χωρών μελών της Ένωσης και χωρών εκτός Ένωσης. Αυτό νομίζω πρέπει να το διερευνήσουμε ακόμη περισσότερο. Η κυρία Χέρση είναι η επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια γιατί κάποια από αυτά που άκουσα πραγματικά με έκανα να θέλω να πάρω το μικρόφωνο. Σίγουρα, όταν μιλάμε για την ε, εμπορία ανθρώπων, πολλές φορές ε, ακούμε συχνά το όνομα μάλλον των Ρωμά, ότι είναι αυτοί που πέφτουν θύματα, αλλά είναι και οι θύτες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να εντοπίσουμε όλα αυτά βέβαια σε μία μόνο ομάδα. Σίγουρα πρέπει να μιλήσουμε για τους Ρωμά, αλλά να μην ε, λέμε ότι είναι μια ομάδα ξεχωριστή, ε, δεν έχουν την ίδια αξία με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους Ρωμά στη συζήτηση που τους αφορά, στη συζήτηση που γίνεται για αυτούς. Στη Σουηδία το ξεχνάμε. Ξεχνάμε να συμπεριλάβουμε τους ίδιους τους Ρωμά στις συζητήσεις μας. Στις συζητήσεις που κάνουμε εμείς για τη στρατηγική για τους Ρωμά. Ο Πρόεδρος. Ακούστε, έχουν υποβληθεί κάποια ερωτήματα. Θα πρότεινα όλοι οι φορείς που εκπροσωπούνται σήμερα σε αυτή τη συζήτηση, το UNDP, η Παγκοσμία Τράπεζα, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, να απαντήσουν με τη γραπτή διαδικασία στα μέλη, στους βουλευτές οι οποίοι υπέβαλαν συγκεκριμένα ερωτήματα και ζητούν απαντήσεις. Γιατί το λέω αυτό. Δυστυχώς δεν μπορώ να διαθέσω άλλο χρόνο για αυτή τη συζήτηση. Διότι πρέπει να βιαστούμε, έχουμε ένα ακόμη ε, σημείο στη μέση διάταξη και στις 12 προβλέπονται οι ψηφοφορίες. Έχουμε ήδη την κυρία Λεμπάγη εδώ, που είναι Γενική Διευθύντρια Δικαιοσύνης και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κοινή συζήτηση που έχουμε στην ημερήσια διάταξη για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πάντω έχει παρουσιάσει την ανακοίνωσή της ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα νέο πλαίσιο για την ε, ε, στρατική ένταξη στον Ρωμά. Και στις επόμενες συναντήσεις της Επιτροπής μας ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε εκ νέου αυτό το πολύ λεπτό ζήτημα που έχει να κάνει με τους Ρωμά και συγκεκριμένα με την κατάστασή τους σε 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτέλεσαν και αντικείμενο αυτής της έρευνας και τις παρουσίες που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Οπότε εδώ θα κλείσω με αυτό το σημείο και θα περάσω στο επόμενο σημείο τη μετσιά διάταξη, που είναι η κοινή συζήτηση για το θέμα τη προστασία δεδομένων. Άρα έχουμε το σημείο 11, προστασία των φυσικών προσώπων αντί της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Με εισηγητή, τον συνάδελφό μα, Γιάν Άλμπρεχτ. Έχουμε και το σημείο 12 όμω προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνουν ή επεξεργάζονται οι αρμόδιε αρχέ για το σκοπό τη πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση ή δίωξη αξιόπινων πράξεων ή εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η συγκητής εδώ αυτων η εδω ειναι ο συναδελφο μα δημητρη Ντρούτσα. Θα έχουμε λοιπόν μια κοινή συζήτηση για τα επόμενα 35 λεπτά. Σύντομοι να είστε παρακαλώ και στις παρουσιάσεις σας οι εισηγητές και στα σχόλιά σας οι υπόλοιποι. Για την προσωπία ε, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ στις ΙΠΑ τον Μάρτιο Είχαμε και ένα workshop για την προστασία των δεδομένων πριν από δύο μέρες. Ε, μας έχουν ήδη δώσει αυτά τα δύο ε, συμβάντα ε, πολλά στοιχεία Έχουμε λοιπόν ήδη εφόδια για να συζητήσουμε σήμερα με τα λόγου γνώσεως τα θέματα της προστασίας δεδομένων. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τον κύριο Άλμπερχτ, μετά τον κύριο Δρούτσα και μετά ενδεχομένως θα ήθελα να κάνουν σύντομες δηλώσεις ε, το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Παρακαλώ κύριο Άλμπερχτ να ξεκινήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω και την δυνατότητα που μας δίνετε εδώ να συζητήσουμε αυτό το μεταρρυθμιστικό πακέτο. Έχουμε ενώπιον μας δύο προτάσεις. Όπως είπατε, έχουμε και την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στα τέλη Ιανουαρίου. Εδώ και κάποιες ε, μήνες λοιπόν ε, συνεργαζόμαστε εντατικά με σκιώδες εισηγητές και εισηγητές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την βασική οδηγία η οποία μας κατατέθηκε, όχι μόνο με τους κοιόδους εισηγητές, αλλά και με τους ε, εισηγητές ε, των ε, επιτροπών που γνωμοδοτούν και με τον κύριο Κέλλη. Και θεωρώ ότι έχουμε σημειώσει ήδη καλή πρόοδο. σε τεχνικές συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε συμφωνήσει επί των βασικών αρχών για τα δικαιώματα των ατόμων. Έχουμε εξετάσει όλα αυτά τα ζητήματα και ασφαλώς εκεί βρίσκεται και ο πυρήνας της νομοθεσίας για το ποιο θα είναι το βασικό οικοδόμημα που θέλουμε να ρυθμίσουμε νομοθετικά στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν τη βάση στην οδηγία του 95. Ακολουθούμε λοιπόν τις αρχές που ορίζονται εκεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζεται και αφετέρου την ελεύθερη κυκλοφορία ε, δεδομένων ε, αναφορικά με άτομα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πολλά έχουν ρυθμιστεί σωστά, έχουν ανακύψει και πάρα πολύ, πολλά ερωτήματα. Έχουμε συνεργαστεί με τους κοιόδους συζητητές αυτά τα θέματα και με τους άλλους συζητητές και υπάρχουν πολλά λοιπόν ζητήματα στα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες ε, ρυθμίσεις. και για τους καταναλωτές και για τη διοίκηση και για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς διατυπώσεις. Θα ψάξουμε να βρούμε τις σωστές προτάσεις μέχρι το θερινό διάλειμμα και μετά το θερινό διάλειμμα, από Σεπτέμβριο πλέον, θα συνεργαστούμε για τα περαιτέρω εκκρεμή ζητήματα, τα οποία ενδεχομένω να πρέπει να συζητηθούν πιο ενδελεχώ. Ε, αυτά είναι θέματα τα οποία ίσως ε, οφείλονται και σε διάσταση απόψεων μεταξύ ημών. Νομίζω ότι έχουμε καλή ε, δυνατότητα, αν συνεχίσουμε τις εργασίες με τον ίδιο ρυθμό, μέχρι τα τέλη του έτους εδώ στην Επιτροπή αλλά και στο Κοινοβούλιο να βρούμε μια κοινή θέση και με την Επιτροπή ΙΜΚΟ και με την Επιτροπή ΙΤΡΕ αλλά και ιδιαίτερως με την Επιτροπή Απασχόλησης και με την Επιτροπή Οικονομικών ε, Θεμάτων που γνωμοδοτούν και αυτές. Ελπίζω να τηρήσουμε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα αυτό. Έχουν προβλεφθεί πολλές συναντήσεις και είναι στενό το χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπεται με τους ε, σκιώδεις. Προχτές είχαμε ένα ενδελεχέστατο εργαστήρι που διοργανώθηκε. 300 συμμετέχοντες. Είναι πολύ έντονο το ενδιαφέρον που εκφράζουν και εξωτερικοί φορείς από την έρευνα, την ανάπτυξη, την οικονομία, από τις ομάδες πίεσης, από την κοινωνία των πολιτών. Όλοι θέλουν να βρεθεί μια σωστή ρύθμιση η οποία θα αποτυπώνει όλες τις πτυχές. Και αυτό το εργαστήρι ήταν μεγάλη επιτυχία, θεωρώ. Πολλές οι εντυπώσεις που συλλέξαμε. Και για τη σημερινή συζήτηση συμφωνώ με τον κύριο Δημήτριο Δρούτσα ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε εκ νέου το συνολικό πακέτο και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της υφιστάμενης οδηγίας. Αυτό ως τώρα χρονικά δεν το καταφέραμε. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη λοιπόν και αυτές οι πτυχές και το τι θα κάνουμε με το συνολικό πακέτο. Εμείς συμφωνούμε από πλευράς εισηγητών και σκιωδών ότι το συνολικό αυτό πακέτο, αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να ολοκληρωθεί στην τρέχουσα θητεία. Βλέπουμε ότι στο βασικό κανονισμό είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι συνηγορούν προς την άποψη αυτή. Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες ελπίζουμε να καταφέρουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας προκειμένου να ξεκινήσουμε να διαπραγματεύσουμε το Συμβούλιο του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τρούτσας τώρα να μας μιλήσει, ο οποίος είναι υπεύθυνο για την ε, δεύτερη εκθέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και θα είμαι πραγματικά σύντομος, καθότι πραγματικά όλο το πακέτο έτσι θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ως πακέτο, αυτό που είπε ο Γιάνν Άλμπρεχτ. Και Επίσης για την οδηγία θέλουμε να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Να διευκρινίσω ότι υπήρξε κάποια απογοήτευση ε, σε ό,τι αφορά την ε, απόφαση να διαιρεθούν το κομμάτι για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε διάφορα τμήματα και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με την, το επίπεδο προστασίας που παρέχει μια οδηγία, ένας κανονισμός. Αλλά όπως και να έχει, εξακολουθεί να αποτελεί ένα πακέτο και σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά ως πακέτο θα το αντιμετωπίσουμε με τον Γιάννη Αλμπρέχ. Προσπαθούμε να δουλεύουμε παράλληλα για τις συζητήσεις ε, για τον κανονισμό και για την οδηγία και οι τεχνικές συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ξεκινήσουν για την οδηγία και υπό την Προεδρία του Συμβουλίου θα γίνουν και άλλε συναντήσει με τον ακαδημαϊκό κόσμο, με τι εθνικέ αρχέ, με την κοινωνία των πολιτών και εμεί και οι σκιώτε θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να συντονίσουμε τι σχετικέ ημερομηνίε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οδηγία, να πω ότι ελπίζουμε η εφαρμογή της να οδηγήσει στην περαιτέρω ενίσχυση των ζητημάτων αστυνομικής συνεργασίας και δικαστικής συνεργασία, ιδιαιτέρως συμπεριλαμβάνοντας ε, την επεξεργασία εγχώριων δεδομένων για να βελτιωθεί η νομική βεβαιότητα για τις αρμόδιες αρχές σε ό,τι αφορά αυτή την δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα και την αστυνομική συνεργασία. Εν συντομία τώρα λίγα λόγια για το περιεχόμενο της οδηγίας, χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Ορίζει τους κανόνες που έχουν να κάνουν με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε ό,τι αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό, την ανείχνευση, την εκτέλεση ποιητικών αδικημάτων και θέτει το διτό στόχο της οδηγίας που είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ελευθερία των φυσικών ατόμων και ιδιαίτερα το δικαίωμα προσωπικών δεδομένων όπου θέλουμε υψηλό επίπεδο ασφάλειας και την διασφάλιση ε, ανταλλαγής τέτοιων δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο σημεία θα ήθελα να τονίσω, τα οποία θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Καταρχάς, οι διατάξεις για τη δυνατότητα μεταφοράς ε, δεδομένων σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς. Εδώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο εξής. Ε οι συνθήκες, οι όροι μεταφοράς θα πρέπει να είναι αρκετά αυστηροί. Και επίσης σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του Εθνικού Φορέα για τη μεταφορά των δεδομένων, θα πρέπει να προσέξουμε να μην είναι περιορισμένε. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη χρηματοδότηση επαρκή. Πού να τονίσω ότι ο βασικός μας στόχος ασφαλώς είναι να διασφαλίσουμε υψηλού επίπεδου και καλής ποιότητας νομοθεσία, η οποία θα αντέξει και στο πέρασμα του χρόνου. Νομίζω ότι και αυτό αποτελεί μια σημαντική πτυχή, την οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη, ότι οι διαδικασίες, οι εξελίξεις, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι πάρα πολύ γρήγορες. Θα πρέπει λοιπόν να αντέξει στο χρόνο το πακέτο το οποίο θα συμφωνήσουμε και ασφαλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την πλήρη προστασία των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών μας. Και επιτρέψτε μου, το έχω πει αυτό και στο παρελθόν, επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι πεπισμένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα πρέπει να διατηρηθεί ιδιαίτερα σε καιρού που στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδείξουμε ειλικρίνεια σε μία περίοδο που έχει χάσει το ειδικό της βάρος και την επιρροή της σε διεθνές προσκήνιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η πρόταση και το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν μια πραγματικά καλή βάση. Και πάλι δράτω της ευκαιρίας για να συγχαρώ την Επιτροπή για το έργο της. Θα ήθελα όμως ένα σημείο να θίξω, να μην επιτρέψουμε οι διατάξεις που προβλέπονται να αποδυναμωθούν στις περαιτέρω συζητήσει με τα κρατημέλη. Αυτό να μας απασχολήσει και ασφαλώς προσβλέπω στη συνεργασία με όλους τους κοιόδης και όλους τους άλλους συναδέλφους έχοντας κατά νου και τη συνεργασία με τους άλλους, τα άλλα όργανα, με τα εθνικά κοινοβούλια, με την κοινωνία των πολιτών, με πάντα από στόχο την επίτευξη της καλύτερη δυνατή ε, νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές. Ποιοι θέλουν το λόγο, πρώτα απ' όλα αρισκιώδης βέβαια. Και μετά θα ακούσουμε την αντίδραση της Κομισιόν και του Συμβουλίου. και της κυρίας Λεμπάγη βέβαια. Και θα κλείσουμε με την ε, σύντομη ε, δευτερολογία των εισηγητών. Παραλαμβάνω, έχουμε πληροψηφοφορίες μετά, στις 12. Ο κύριος Άλβαρ Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ο κύριος Άλβαρο να μην ξεχνάμε στο πλαίσιο αυτό να ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βουλευτές. Έχουμε κάποια σημεία κριτικής και στο σημείο αυτό θα ε, παρουσιάσουμε τη δική μας προσωπική άποψη και αυτό ε, εξαρτάται φυσικά από το που προέρχεται και ο καθένας, αλλά με πάσα ειλικρίνεια θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι απλό να διαμορφώσουμε ένα πακέτο που να ικανοποιεί όλους. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εντατική της εργασία που μας υπέβαλε και το έργο της που μας παρουσίασε αρχές του έτους. Ο κανονισμός επιφέρει μια βασική αλλαγή σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παντού ε, την αρχή του χώρου αγοράς. Δεν χρειάζεται μία εταιρεία να έχει έδρα στην Ευρώπη για να υπόκειται στο σχετικό δίκαιο. Όχι, φτάνει να απευθύνεται σε πελάτες στην Ευρώπη. Με το τομέα αυτό λοιπόν πετύχαμε κάτι το οποίο εδώ και καιρό συζητούσαμε. Κάναμε ένα πρώτο βήμα λοιπόν στην Προ την προστασία δεδομένων ανεξαρτήτως τόπου για τον Ευρωπαίο πολίτη. Ενδιαφέρουσε άλλε ε, αρχές είναι το privacy by default, privacy by design. Θα πρέπει όλα αυτά να κοιτάξουμε πώ διαμορφώνονται. Σε ό,τι αφορά το privacy by design, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν ε, προδιαγραφές ασφαλείας που θα πρέπει να τηρούνται στην αγορά σε ό,τι αφορά ε, διαγωνισμούς και θα πρέπει να ομολογήσω θα πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το effect 2.0 δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η βελτίωση που υπάρχει σε σχέση με την προηγούμενη αρχή διαγραφής. Ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσον να υπάρχει ε, ένα δικαίωμα να ξεχαστεί κανείς πλήρως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είναι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες έχει μειωθεί η γραφειοκρατία. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές στην οδηγία. Θα πρέπει να σας πω ότι οι σχέσεις σε ό,τι αφορά την, ε, τον υπεύθυνο προστασία των δεδομένων στο σημείο αυτό έχουν επισέλθει κάποια καινούργια στοιχεία λοιπόν και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε το τι αλλάζει πραγματικά. Το One Stop Shop ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός ε, consistency, γιατί ε, το data shopping ε, νομίζω ότι έχει τεράστιες επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιμετωπίζουμε, θα αντιμετωπίσουν οι αρχές ε, προστασίας δεδομένων τεράστιες προκλήσεις σε ό,τι αφορά το αυξημένο προσωπικό που θα χρειαστούν. Νομίζω λοιπόν ότι η, πρακτική, η πράξη θα πρέπει να δημορφωθεί με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει υπερβολικά τις ε, τοπικές αρχές. Και νομίζω ότι στο πλαίσιο των σκιωδών θα πρέπει να συζητήσουμε με τους ε, συγητές ε, αν οι εξαιρέσεις όπως διαμορφώνονται που ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού μήπως θα πρέπει να οριστούν πιο στενά Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά κοιτάξτε πώς να κοιτάξουμε 100 άρθρα σε δύο λεπτά. Και για να ολοκληρώσω, νομίζω ότι ενδιαφέρον θα ήταν αν μπορούσαμε να κάνουμε μία αναφορά και στο κοινωνικότερο πλαίσιο, πώς τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται αξιοποιούνται και τέλος τέλος, γιατί βλέπω ότι είναι και νευρικός ο Πρόεδρος, να αναρωτηθούμε γιατί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρούνται. Και μήπως θα έπρεπε να διευρυνθεί ο κανονισμός και για τα ευρωπαϊκά αυτοθεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, υπομονή σας. Ευχαριστώ κύριε Φως για τρία λεπτά. Ähm, ευχαριστώ πολύ. Να μην επαναλάβω όλα όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητέ, αλλά θεωρώ ότι είναι αξιέπαινο το γεγονό ότι υπάρχει καλή σχέση μεταξύ των εισηγητών και ιδιαίτερω ε, μεταξύ του Γιάνν Φιλιππ Άλμπρεχτ και του Δημήτρη Βρούτσα. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερω ε, που σε ό,τι αφορά το πακέτο προστασία των δεδομένων ε, καθόμαστε και σκεφτόμαστε τι θα πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τη γενικότερη κατεύθυνση της νομικής πράξης και το θέμα της συμπερίληψης του δημοσίου τομέα, το θέμα του τι εννοείται ε, με τα αρχεία δεδομένων, όλα αυτά τα αναφέρει και ο κανονισμός. Θα πρέπει να κάτσουμε να κοιτάξουμε τον κανονισμό προκειμένου να διαμορφωθεί ε, με τρόπο εφαρμόσιμο και πρακτικό στην πράξη θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τις ημερομηνίε που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά στο διάλογο αυτό φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές παρανοήσεις, πάρα πολλές ε, διαφορές μεταξύ της ε, πράξης και της πρόθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο σημείο λοιπόν αυτό θα πρέπει να εξαλειφθούν αυτές οι διάφορες και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο direct marketing, balance of interest clause. Εδώ υπάρχει ασάφεια πρέπει να διευκρινιστούν αυτά νομικά. Τώρα, αυτό αφορά πάρα πολλά σημεία όπου έχω την αίσθηση ότι δεν διευκρινίζονται απαραίτητα όσο πρέπει τα πράγματα. Ισχύει για παράδειγμα on and offline, τι ισχύει για το θέμα του online, το δικαίωμα right to be forgotten, όπως αναφέρατε, μπορεί να μην έχει τόσο πολύ νόημα να ισχύει, για παράδειγμα, αυτή η υποχρέωση για νοσοκομεία, για ασφάλειες. Υπάρχουν κάποιοι τομείς, λοιπόν, που θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε τι θα γίνει στην πράξη και πώς. Σε αυτά θα ήθελα να περιοριστώ, γιατί τα σημεία που ανέφερε και ο κύριος Άλβαρο, αλλά και οι ήταν σωστά. Χρειάζεται πιο μεγάλη σαφήνεια, γιατί υπάρχουν, ε, υπάρχει διαίρεση απόψεων. Το συζητήσαμε και στο εργαστήρι. Νομίζω ότι σε σωστό δρόμο βρισκόμαστε και ελπίζω να μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, γιατί η περιπλοκότητα του θέματος αυτού είναι τόσο μεγάλη που πρέπει να έχουμε τον κατάλληλο χρόνο για να συζητήσουμε επαρκώς όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κέλλη, συγκεκριτής από την Επιτροπή Ήτρε, αν θα θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, γι' αυτό θα είμαι σύντομο. Το εκτιμώ ότι μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω. Σημαντικότατο θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εφαρμόζουμε αυτό που θέσπισε και το 95 πανστατικές αλλαγές όσον αφορά την προστασία των δεδομένων ανάπτυξη τεχνολογίας που έλαβε χώρα έκτοτε. Χρειαζόταν λοιπόν κανονισμός. Τονίζω, κανονισμός δεν αρκεί οδηγία. Χρειαζόμαστε κανονισμό και καλό. Θα συζητήσουμε κατά πώς θα ακολουθήσουμε το άρθρο 50 του 49. Ούτως ή άλλως προσβλέπω συνεργασία με τον εισηγητή, τον κύριο Άλμπρεκτ. Ήδη συναντηθήκαμε πανελειμμένα. Μου θυμίζει ένα ρητό στη γλώσσα μου. Οπότε λέει, δεν, ε, ισχύσαν τη ενώση με λίγα λόγια. Μπορεί να έχει ό,τι οι δεξιότητε θε, αν δεν υπάρχει συνεργασία, δεν θα υπάρξει πρόοδο. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε για να έχουμε τον καλύτερο δυνατό κανονισμό για να προστατεύεται το άτομο και να επιτρέπουμε και σε επιχειρήσεις να αναπτύσσουν και να προωθούν τη διαδικασία της ε, πρόσβασης των επαφών μέσω διαδικτύου online. Τέλος. Έκανε αξιολόγηση σε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν αρκετά πλήρης. Αλλά δεν αρκεί, κατά την άποψή μου. Θα πρέπει το τμήμα του Κοινοβουλίου που είναι υπεύθυνο εξολόγηση αντιχτύπου θα πρέπει να κάνει και αυτό για μας μια μελέτη αντιχτύπου και έτσι θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε. Αυτό ήθελα να σας ζητήσω σήμερα. Ευχαριστώ που υπήρξατε σύντομο. Κυρία Ένστ για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομη. καταρχά να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα του συζητητέ. Είναι σχεδόν, τι να πω, εκπληκτικό. Κοιτώντα το συνολικό πακέτο των εκδηλώσεων, συναντήσεων, συζητήσεων, εργαστηρίων, είναι σημαντικό που γίνεται αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Είναι σημαντικό να ρωτάμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς κατέληξε στα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε. Την ευχαριστήσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα λοιπόν που μας απασχολεί ποιο είναι να υπάρχει μια συνολική προσέγγιση, ένα συνολικό πακέτο υψηλής ε, δεσμευσιμότητας, ε, υψηλής διαφάνειας και για τον εμπλεκόμενο πολίτη κυρίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Χρειαζόμαστε τεχνική ουδετερότητα, χρειαζόμαστε κατάλληλο επίπεδο σε όλα τα κατημέλη και φυσικά δεν μπορεί να περιοριστεί το επίπεδο σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά θετικά στοιχεία τα οποία αναφέραμε, η ενίσχυση του υπεύθυνου και τα προσωπικά δεδομένα ανά κράτος μέλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, με απασχολεί ιδιαίτερα και η ειδική συμπερίληψη παιδιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για μένα. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι εκκρεμή και θα πρέπει να συζητηθούν. Για παράδειγμα, το πεδίο εφαρμογή αναφέρθηκε ήδη. Είναι κάπω ατυχέ το γεγονό ότι κάποιοι τομεί εξαιρούνται, όπω η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα. Ε, πολλά θα πρέπει να διευκρινιστούν και πολλοί ορισμοί. Διαπιστώνω ότι κάποια πράγματα τα οποία στην αρχή μου φαινόντουσαν απλά δεν είναι απλά, για παράδειγμα, η πρώτος ο ορισμός, αυτό το δικαίωμα να ξεχαστεί κανείς, το profiling. Και εδώ θεωρώ ότι κάποια πράγματα δεν μπορεί να παραμένουν ως έχουν. Και ένα μεγάλο πρόβλημα έχω επίσης με το ε, delegated acts, με τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε πού θα πρέπει να συμπεριληφθούν και πού όχι. Αυτό φυσικά μόνο βαθμιαία μπορεί να αποφασιστεί ανάλογα με την κατάσταση. Για την οδηγία τώρα, για την προστασία των δεδομένων, για τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, θεωρώ ότι είναι μάλλον επισκιασμένες αυτές οι δύο αρχές ως τώρα. Και στην οδηγία προκύπτουν μια σειρά προβλημάτων που θα πρέπει να συζητήσουμε. Θεωρώ ότι όταν μια οδηγία αναφέρει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το αναφέρει με πολύ σαφή διατύπωση, γιατί είμαι κάπως διστακτική σε ό,τι αφορά την εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο, σε πολλά θέματα. Και νομίζω ότι πολλά ε, τέτοια θέματα θα πρέπει να χτενίσουμε στο άρθρο 10, στο άρθρο 11, ε, διατάξεις laissez-faire, αλλά και σε άλλους τομείς. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε εν συντομία και σίγουρα στις συναντήσεις με τους συζητητές θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Πάντα σε συνάρτηση και με τον κανονισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ε, κυρία Χέντ, τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να πω μερικά λόγια για την έκθεση Albrecht. Είναι το πληρέστερο νομοθέτημα αυτής της θητείας. Καλύπτει πολλούς τομείς. Άρα είναι σημαντικό να μην φυστούμε χρόνο για να κάνουμε σωστή δουλειά. Προτείνονται κάποια πράγματα την προστασία των δεδομένων. Έχουμε τεχνικές εξελίξεις μετά το 1995 άλλαξαν πολλά. Και συμπεριλαμβάνονται στην Πρωθυπουργική Επιτροπή. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται η επιλογή ε, κανονισμού και όχι οδηγία. Όταν μιλάμε για στοιχεία για ασθενεί όμω, ίσως εκεί μπορούν να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα προστασία ε, και εκτός κανονισμού. Ίσως έτσι ε, έχουμε ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας, αλλά χαμηλότερο. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης. Δεν θα πρέπει να περικοπεί. Και τι γίνεται με τις εξαιρέσεις για την επεξεργασία των δεδομένων, για δημοσιογράφους, Φερρυπίν. Πρέπει να το προσέξουμε. Και σύγκρουση μεταξύ διαφανής και προστασίας των δεδομένων πρέπει να εξεταστεί η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων χρησιμοποιείται σε δικαιολογία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη παροχή πληροφοριών για την υποστήριξη στον αγροτικό τομέα. Ελπίζω ότι αυτός ο κανονισμός δεν θα χάσει τη μάχη για τους καταναλωτές, για περισσότερες πληροφορίες. Είμαστε ε, ε, ε, Πρέπει να υπάρχει ανοιχτή προσέγγιση και διαφάνεια όπως στη χώρα μου. Ελπίζω αυτό να το επεξεργαστούμε εγκαίρω και διαφανώ. Oh, ε, κυρία Ινβέλτ. Είναι εδώ. Όχι. Λυπούμε. Δεν τη ζήτησε το λόγο. Αλλά απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Ας ακούσουμε τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και μετά πάμε στους εισηγητές για να κλείσουμε. Η κυρία Λεμπάη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι ενθαρρύνομαι τα μάλα από αυτά που άκουσα. Είναι μια δέσμη προτάσεων που και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν κοινό στόχο. Υψηλό επίπεδο προστασία δεδομένων δηλαδή στην Ευρώπη. Οι προτάσεις που κάναμε πράγματι είναι πολύ φιλόδοξες. Είναι μια δέσμη προτάσεων. Και βασιζόμαστε κατά πολύ στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο ώστε να εξακολουθήσει αυτή η προσέγγιση. Θα αντιμετωπίσετε κι εσείς όπως και εμείς ε, θέση διαφόρων πάρα πολλών τεχνικών σημείων από το Συμβούλιο. Πρέπει να έχουμε υπόψη όμως τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε υψηλό επίπεδο, υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους πολίτες. Σημαντικότατο ζήτημα. Πολλά στοιχεία των προτάσεών μας έχουν αυτό το στόχο. Πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες που θα συζητηθούν, αυτό είναι ο σκοπό μας, που πρέπει να παραμείνει υπόψη μας. Δεύτερο στοιχείο των προτάσεων. Απλούστευση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι υψηλό βαθμός προστασίας δεδομένων μπορεί να συνδυαστεί με ανάπτυξη, με συνεισφορά στην ανάπτυξη. Δεν πιστεύουμε ότι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων δυσκολεύει ε, τη ζωή των επιχειρήσεων. Καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες σχετικά. Έκαναμε διάφορες προτάσεις που εξαιρούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραδείγματος χάρη από τις διάφορες ε, λεπτομέρειες για την εφαρμογή. Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε τυχόν καλές ιδέες στον τομέα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έτσι περαιτέρω. Ε, τρίτο στοιχείο. Ε, σωστή εφαρμογή με τους διάφορους φορείς συνεργαζόμαστε για να δοκιμάσουμε, να δούμε κατά πόσο ε, μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιε θα είναι οι συνέπειες για τους πόρους, για τους φορείς που εφαρμόσουν τα μέτρα. Ζητήσαμε τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν το ότι οι αρμόδιοι φορείς θα έχουν τους αναγκαίους πόρους, στελέχωση, οικονομικούς πόρους. Κρισίμου σημασίας. Τέταρτο στοιχείο και χαίρομαι για αυτά που μας είπαν οι συγγητές πάνω σε αυτό. Πρέπει αυτή η δέσμη μέτρων παραμείνει συνεκτική. Κανονισμός και οδηγία. Είναι σημαντικότατο. Διότι η αρχή για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να εφαρμόζεται και στους δύο τομείς. Στον αστυνομικό τομέα υπάρχουν παρεκκλήσεις, εξαιρέσεις. Κανονικό, συνηθισμένο αυτό, το έχουμε υπόψη μας Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος πως στόχος και των δύο συγητών είναι να παραμείνει ενία η δέσμη μέτρων. Χρονισμός, τελευταίο σημείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ φιλόδοξη. Και από την πλευρά σας παρομοίως. Θέλω αυτό το πακέτο να υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντικό για τους πολίτες και για τις επιχείρησεις. Ό,τι βοήθεια μπορούμε να παράσχουμε με τα χαράς να το κάνουμε. Η συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου πηγαίνει πάρα πολύ καλά και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή και να την αυξήσουμε μάλιστα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Λεμπάιλ για την προσπάθεια που κάνατε για να απαντήσετε στα περιπλοκότατα ζητήματα αποφεύγοντας τεχνικές λεπτομέρειες. Παρακαλώ, ησυχία, ησυχία όσοι μένουν στην αίθουσα. Διανέμονται οι κατάλογοι ψηφοφοριών. Αλλά παρακαλώ, ήσυχα. Αλλιώς δεν τα καταφέρουμε. Το Συμβούλιο, λοιπόν, έχει το λόγο. Θέλει να πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Από πλευρά Συμβουλίου, Πρέπει να πω ότι κάναμε διάφορες συνεδριάσεις με θέμα τις δύο προτάσεις, κυρίως όσον αφορά τον κανονισμό συζητήσαμε εκτενώς για την οδηγία. Το συζητήσαμε σε επίπεδο ομάδων εργασίας και σε ψηλότερο επίπεδο, σε ομάδες εργασίας υψηλού επίπεδου. Έγινε ζωή συζήτηση στο Συμβούλιο, διάφορα ερωτήματα έχουν τεθεί και παρόμοια ζητήματα με αυτά που έθιξαν οι βουλευτές. Είναι θέματα που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι επικρατεί η άποψη στο Συμβούλιο ότι χρειάζεται ενημέρωση οδηγίας του 95 διότι το παρόν πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Χρειαζόμαστε δέσμοι μέτρων που ανταποκρίνεται στη δοκιμασία του χρόνου. Θέλουμε υψηλά επίπεδα προστασίας. Συζητήσαμε το πεδίο εφαρμογή, τις νέες αρχές πώς θα εφαρμοστούν πρακτικά το διοικητικό άχθος, η δομή των νομικών πράξεων, δημόσιος, ιδιωτικός τομέας, πώς θα ταιριάξουν. Αυτά είναι θέματα παρόμοια με αυτά που εξέφρασαν τα μέλη σήμερα. Σημαντικότατο ζήτημα. Μας περιμένει πολλή δουλειά στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Συμβούλιο για τα σχόλια. Και πάλι να στραφούμε προς τους συζητητές και πάλι όμως να επαναλαμβώ ότι όσοι είναι στην αίθουσα παρακαλώ να μην κάνουν κατευθείαν συζητήσει. Ξέρω ότι σας μοιράσαμε τους κατάλογους ε, ψηφοφορίας. Σας παρακαλώ ησυχία όμως. Debate which is the final part, the conclusions by the rapporteurs, Mr. Albrecht. Ο κύριος Albrecht. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους του συναδέλφους για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ανταλλαγή απόψεων για το πακέτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, να το αντιμετωπίσουμε ως ένα ενιαίο πακέτο, το οποίο από κοινού θα πρέπει να εξετάσουμε. Να επαναλάβω, έχοντας ακούσει και αυτά που είπε το Συμβουλίο, ανυπομονώ ιδιαίτερος. Να γίνουν και οι πρώτοι μας ανεπίσημες συναντήσεις να ακούσουμε και την άποψη του Συμβουλίου για το ποια θέματα του απασχολούν ιδιαίτερα, γιατί δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε τριμερείς διαλόγους από εντελώς διαφορετικά σημεία εκκίνησης, ίσως να έχουμε παρόμοιες ιδέες για το πώς θα βελτιωθούν οι προτάσεις. Και μια τελευταία κουβέντα για τη συνεργασία εδώ. Χαίρομαι που ο κύριος Κέλλη από την Επιτροπή Ήτρε ε, παρευρίσκεται. Θα συνεργαστούμε και με την Επιτροπή ΕΜΚΟ και ελπίζουμε να βρούμε λύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα, για το ποιος ε, κανόνας θα πρέπει να εφαρμοστεί. Νομίζω όμως ότι θα είναι καλή συνεργασία και θα βρούμε λύσεις. Και ελπίζω την άλλη φορά που θα βρεθούμε εδώ να έχουμε μία πρώτη ιδέα για το πού θέλουμε να γίνουμε αλλαγές, ποια ζητήματα, σε ποια ζητήματα συγκλίνουν οι απόψει μας και σε ποια όχι. Μα σας παρακαλώ διακόπτει ο Πρόεδρος. Τι γίνεται. Μιλάει βουλευτή. Σας παρακαλώ. Δεν θέλω κατευθείαν συζητήσει. Κύριε Άλμπρεχτ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι όλοι οι σκιώδει και εγώ πάντα είμαστε αντιτεθειμένοι να συζητήσουμε μαζί σας ε, ενδεχόμενα θέματα τα οποία σας απασχολούν και τα οποία θα ανακύψουν στις συναντήσεις. Ε, φυσικά προγραμματίζονται διάφορες συναντήσεις, όλα με τη σειρά τους ασφαλώς. Αν χρειαστεί, σας παρακαλώ να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Άλμπρεχτ και τώρα κύριε Στρούτσας για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους σας για τις παρεμβάσεις σας, ιδιαίτερα για το πνεύμα συνεργασίας που επιδείξατε. Και είμαι πραγματικά πεπισμένος ότι το όλο πακέτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας πολιτικής, ένας από τα πιο σημαντικά ζητήματα μάλιστα της ε, υπόλοιπης Και πάλι να σας καλέσω όλους να έρχεστε σε επαφή με εμάς τους εισηγητές και τους κοιόδες εισηγητές ασφαλώς, αλλά και τους ε, υπόλοιπους βουλευτές, τα υπόλοιπα μέλη. Να μας πείτε ποιες είναι οι ιδέες σας, γιατί τονίζω εκ νέου ότι το πακέτο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφορά τα δικαιώματα του πολίτη, αυτόν εκπροσωπούμε εδώ και θα πρέπει λοιπόν να τα πάρουμε όλα αυτά στα σοβαρά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρο, Όλα αυτά λοιπόν ολοκληρώνουν τη συζήτηση αυτή, την κοινή συζήτηση σε ό,τι αφορά τα θέματα προστασία των δεδομένων. Και τώρα ξεκινάει η ψηφοφορία. Να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι? Τις ηλεκτρονικές σας κάρτες, μην ξεχνάτε, έχουμε ένα λεπτό πριν ξεκινήσουμε ψηφοφορίες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 Dear colleagues. Συνάδελφοι. Get ready. Get ready to go. Έτοιμοι. Έχετε τις κάρτες σας. Πριν από την ψηφοφορία. Dear colleagues, ladies and gentlemen, take your... Σας παρακαλώ καθίστε συνάδελφοι. Συγκεντρωθείτε στην ψηφοφορία. Δεν πρόκειται να είναι εύκολη. Έχουμε κάποιες δυσκολίες σε ό,τι αφορά τις ψηφοφορίες και να σας επιστήσω την προσοχή σε κάποιες εξ αυτών. Καταρχάς, χτες έγινε συνάντηση των συντονιστών, εξετάσαμε το σύνολο της ατζέντα, τα συνηθισμένα, αλλά έγινε και μία συζήτηση για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για τις ε, αποστολές στο εξωτερικό της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Έγινε μια συζήτηση για την αντιπροσωπεία που προβλέπεται να αποσταλεί στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, για μια έκθεση που δόθηκε στην Επιτροπή μας ε, τον Φεβρουάριο για την ε, κατάσταση στην Ουγγαρία. Η Επιτροπή μας ήταν η Καθαήλ Αρμόδια, η οποία θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, να ολοκληρωθεί για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρόταση αποστολής στην Ουγγαρία, αλλά λόγω έλλειψης ε, θέσεων βάσει των αποφάσεων που είχαν γίνει και για άλλες αποστολές στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έγινε λοιπόν η συζήτηση αυτή για την αποστολή στην Ουγγαρία. Ελήφθη απόφαση να ψηφιστεί η δυνατότητα αποστολής της Επιτροπής μας στην Ουγγαρία, αλλά από ό,τι ακούσαμε ο συνάδελφος ε, κύριος Ταβάρες, ο εισηγητής, ε, θέλει να πάρει το λόγο για να μας διαφωτίσει για το πώς έχει κατάσταση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να πω ότι η αντιπροσωπεία, η αποστολή στην Ουγγαρία στο πλαίσιο της έκθεσης ε, για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωση δεν διακυβεύεται. Μας κάλεσε ο ίδιο ο, Ορμπαν, ο Όρμπαν ε, στο Στρασβούργο να μεταβούμε στην Ουγγαρία. Και όλα τα μέλη της Επιτροπής έχουν ταχθεί υπέρ της αποστολής αυτής. για την αξιολόγηση της κατάστασης στη χώρα αυτή. Προσωπικά συνομίλησα και με τις ηγεσίε των πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο και όλοι είναι υπέρ της αποστολής στην Ουγγαρία. Εκ παραλλήλου υποσχεθήκαμε στην πρώτη τελαγή απόψεων η αποστολή αυτή να επιδείξει ανοιχτό πνεύμα και να έχει και όσο πιο δυνατόν ευρεία σύνθεση. Καταρχάς λοιπόν θέλουμε μία ad hoc αποστολή στην Ουγγαρία, επειδή και η ίδια η έκθεση στο πλαίσιο της οποίας ε, διοργανώνεται η αποστολή αυτή είναι έκθεση ad hoc που έχει ζητήσει η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Επίσης έχει γίνει μια συμφωνία και για τις ημερομηνίε. Νομίζω ότι μίλησα με όλους τους κοιόδης. Σας παρακαλώ ησυχία, λέει ο Πρόεδρος. Όλοι οι σκιώτες εισηγητές από όλες τις πολιτικές ομάδες συμφώνησαν ότι ο Σεπτέμβριος και ιδιαίτερα στην τελευταία εβδομάδα είναι η πλέον κατάλληλη ε, εβδομάδα για την αποστολή στη Βουδαπέστη. Ε, ήρθα σε επαφή με, τον πρόεδρο, με το γραφείο του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου μου, τον κύριο Μάρτιν Σούλτς, και να ενημερώσω την Επιτροπή μας ότι ε, μπορούμε να συζητήσουμε το συντομότερο δυνατόν την αποστολή αυτή, την ad hoc αυτή ε, αποστολή στη Βουδαπέστη. Ενδεχομένως να συζητηθούν αυτά και σήμερα αύριο στην Κύπρο. Άρα θεωρώ ότι είναι μάλλον πρόημο στην παρούσα φάση να συζητηθεί και να ψηφιστεί η αποστολή στην Ουγγαρία εγώ θα έλεγα να σας υποστηρίξουμε εσάς, Πρόεδρε της Επιτροπής μας, να αποστείλετε καταπήγουν έτοιμα προς την διάσκεψη των Προέδρων για να αποφασιστεί ο αριθμός των μελών της αποστολής και μετά θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μετά την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων. Μάλιστα τα ακούσαμε λοιπόν, ε, ακούσαμε την πρόταση του συναδέλφου του εισηγητή κυρίου Ταβάρες που μας υπενθυμίζει ότι η έκθεση αυτή για την Ουγγαρία δεν είναι κάτι το προαιρετικό, είναι υποχρεωτική. Μας την ανέθεσε μάλιστα η σχετική απόφαση της Ολομέλειας, αλλά θα μπορούσαμε να αποφύγουμε ενδεχομένως τώρα την ψηφοφορία υπό τον όρο ότι θα πρέπει να απευθυνθώ εγώ στη διάσκεψη των Προέδρων για να διασφαλίσω ότι θα έχουμε την επιλογή σε ό,τι αφορά τα μέλη της αποστολής. Είχαμε αποφασίσει λοιπόν ε, επ' αυτόν. Δεν ξέρω, συμφωνείτε, έχετε αντιρρήσεις, ενστάσεις. Αν δεν έχετε αντίρρηση, δεν θα γίνει σχετική η ψηφοφορία και θα προχωρήσουμε με τις ψηφοφορίες που αναφέρονται στον κατάλογο ψηφοφοριών τα έχετε μπροστά σας. Καταρχάς, ε, εντολή για τον τριμερή διάλογο προϋπολογισμός 2013. Εισηγητής, ο συνάδελφος Ιακολίνο. Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, λάβετε θέσεις. Δεν θα είναι απλή η ψηφοφορία, ας ε, ε προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 που είναι συμβατή με την συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στη συμβιβαστική. Α, να το ελέγξουμε. Ωραία. Αν θέλετε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη συμβιβαστική 2. Τη συμβιβαστική 2, ηλεκτρονικός έλεγχος. Α, περιμένετε, περιμένετε. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Σας παρακαλώ, για κοιτάξτε. Δύο, δύο περισσεύουν από το ΕΛΚ. Δύο επιπλέον ψηφίζουν για το ΕΛΚ. Εντάξει. Πολύ ωραία. Τώρα. Is it right now? No, no, I have not voted. Now, now they vote. No, no. Ναι, μα συγγνώμη, δεν έχουμε κάνει την ψηφοφορία. Τώρα θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Τώρα, λοιπόν, έναρξη ψηφοφορία για τη συμβιβαστική δύο. Τώρα περισσεύει ένας από τους σοσιαλδημοκράτες και ένας από το ΕΛΚ. Still one S&D. And how does it go? One S&D. One S&D too many. Τώρα περισσεύει ένας από τους σοσιαλδημοκράτες. Για να δούμε. Ποιος ψηφίζει. What do we get? Well, somebody has to take Could anybody from the S&D withdraw the vote? Withdraw? Yes. Now. Μάλιστα. Ωραία. 27 υπέρ, 30 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σεμιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σεμιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, ας το ελέγξουμε. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη συμβαστική 4, παρακαλώ. Now, one EPP too many. One... E Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Μάλιστα. Ωραία. 29 υπέρ 20 κατά εγκρίνεται. Και τώρα, τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε όμως αν θέλετε. Παρακαλώ έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την τροπολογία υπαριθμών 14. Πέρας της ψηφοφορίας. 30 υπέρ 29 κατά. Έγκρινεται. Η 15 όχι, συγγνώμη. Η συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και τώρα Τροπολογία 18 σε δύο τμήματα. Τρία τμήματα, συγγνώμη. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της 18, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές, ας το ελέγξουμε αν θέλετε. Ηλεκτρονικός έλεγχος, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 27 παρακαλώ. Γιατί και στις νομάτες μέσα δεν υπήρχαν σαφήνεια. Για την 27 λοιπόν τώρα να ψηφίσουμε αν θέλετε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 30 υπέρ 28 κατά εγκρίνεται. Και τώρα η 30 παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω. Θέλετε να το ελέγξουμε. Θέλετε να ελέγξουμε την 30. Εντάξει. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία περιθμών 30 παρακαλώ. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. 30 υπέρ 29 κατά εγκρίνεται. Η 31 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Now closed. Πέρας. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Τώρα. Ολοκληρώθηκε η ψηφορία. 48 υπέρ, 5 κατά, 4 αποχές, εγκρίνεται. Μπράβο στον κύριο Γιακολίνο. Now we've got the draft opinion. Περνάμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης για τη συμβατότητα κτλ. Τη συμφωνία κατά τη απομίμηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κατώμερων και Αυστραλία, Καναδά, Ιαπωνία, Κορέα, ε, Μεξικό, Μαρόκ, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ελβετική, Συνομοσπονδία Πολιτειών, με τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο χάρτη των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Δρούτσα, θέλετε να διευκρινίσετε κάποια πράγματα από ό,τι κατάλαβα πριν την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο ψηφοφοριών, έχει τροποποιηθεί σήμερα το πρωί με τη δική μου συνένεση. Θέλω να γίνει και μία ακόμη αλλαγή σε ό,τι αφορά την τροπολογία 37 το ΕΛΚ ζήτησε σε περίπτωση που η τροπολογία 37 εγκριθεί αυτό να έχει ως συνέπεια τα λοιπά τμήματα της συμβιβαστικής τροπολογίας να καταστούν περιτά, να καταπέσουν. Τα βλέπετε στον κατάλογο για αυτά τα τμήματα. Σήμερα το πρωί όταν μου υποβλήθηκε το αίτημα, το δέχτηκα. Και αυτό όχι γιατί επί της ουσίας συμφωνώ. Εδώ ισχύει το αντίθετο. Διαφωνώ. Αλλά είπα ναι, διότι πιστεύω βαθιά στις δημοκρατικές διαδικασίες. Και αν μια πολιτική ομάδα έχει ένα αίτημα, θέλω να το δεχτώ. Έτσι συνηθίζω. Ότι υπήρχαν σοβαρές αντιδράσεις όσον αφορά αυτή την απόφαση με πολύ σωστά επιχειρήματα και γι' αυτό και πάλι λέω ότι πιστεύω ένθερμα στις δημοκρατικές διαδικασίες. Βλέπω ότι περισσότερες πολιτικές ομάδες μάλιστα δεν συμφωνούν με την αλλαγή που συμφωνήσαμε το πρωί και γι' αυτό θα ήθελα ο Πρόεδρος να αποδεχθεί αυτή την αλλαγή που ζητώ, δηλαδή να γίνει ο, ο κατάρρος όπως ήταν πριν, πριν την πρωινή τροπολογία. Με άλλα λόγια, αν η τροπολογία 37 υιοθετηθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι τα τμήματα της συμβαστικής τροπολογίας 7 που γίνονται πλεονασμοί θα ψηφιστούν και στη συμβαστική. Ευχαριστώ κύριε Δρούτσα. Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να βιαστούμε εδώ, διότι προβλέπονται εργασίες μέχρι το 2030, έχουμε ακόμα ψηφοφορία. Προτείνω εκπρόσωπος κάθε ε, ομάδας να εκφράσει τη θέση της. Κύριε Μπουσετήλ. Συμφωνείτε με την πρόταση που έκανε ο κύριος Δούτσας. Κύριε Πρόεδρε, όχι, δεν συμφωνώ και ζητώ να αποφασίσετε. Υπάρχουν διαφορετικά συμπεράσματα που μπορεί να θετήσει η γνωμοδότηση. Μία είναι να συστήσει απόρριψη της άκτα, άλλη λύση είναι να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασκεδάσει τις ανησυχίες που αναφέρονται στην γνωμοδότηση. Αυτά είναι δύο διαφορετικά συμπεράσματα και εξορισμού είναι ε, ασύμβατα. Αν το δεύτερο συμπέρασμα εγκριθεί από εμά σήμερα, είναι σαφές ότι θα επικρατήσει του πρώτου συμπεράσματος που είναι να συσταθεί η απόρριψη. Και γι' αυτό σας ζητώ κύριε Πρόεδρε, αντίθετα με αυτά που μας είπε μόλις τώρα ο συγητής να αποφασίσετε να παραμείνει η ερμηνεία που έχουμε στον κατάλογο ψηφοφοριών δηλαδή εάν η τροπολογία 37 εγκριθεί τότε προφανώς θα καταργήσει το τελικό τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας 7. Δεν για την τροπολογία 37. Αν είναι παραδεκτή είναι το θέμα, διότι υπευλήθη μετά την εκπνοή της προθεσμίας. Σαν τεχνική αλλαγή υπευλήθη. Πιστεύω ότι αλλάζει περισσότερο το περιεχόμενο και είναι ε, και καλυμμένο αυτό και παρουσιάζει τεχνική ε, τροπολογία, ενώ ουσιαστικά τροποποιεί την ουσία. Πρόεδρος, από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η τροπολογία δεν υπευλήθη εκ των υστέρων μετά την προθεσμία. Υπευλήθη από τους προ... πρασίνους σαν προφορική τροπολογία. Σύμφωνα με τους κανόνες. Ας ακούσουμε την κυρία Ιντβελτ. Προσπαθώ να πετύχω συνένεση επί της προτάσεως του κυρίου Δρούτσα. Η κυρία Ιντβελτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς βλέποντας το κείμενο της τροπολογίας 37 Αντίθετα τον κύριο Μπουσετήλ δεν νομίζω ότι είναι ασύμβατη και αν είναι ασύμβατη γιατί ανακαλύφθηκε μόλις σήμερα το πρωί και τέθη από το ΕΛΚ. Δεύτερον, δεν είναι απλή τεχνική προσαρμογή του καταλόγου ψηφοφοριών και είμαι αρκετά εκνευρισμένη παρουσιάστηκε τούτο τρόπος. Παίρνουμε εκατοντάδε ηλεκτρονικά μηνύματα. Πήρε ένα από τη γραμματεία για την τεχνική προσαρμογή του καταλόγου ψηφοφοριών και ανακαλύπτω ότι δεν είναι καθόλου τεχνικό διότι αφορά ακριβώς τον πυρήνα, την καρδιά του ζητήματος. Διότι αν αποδεχτούμε την πρόταση του ΕΛΚ, που δεν είναι τεχνικής φύσης, αλλά άκρο πολιτική, τότε αντίθετα με αυτά που ο κύριος Δρούτσας και, και συγγνώμη που διαφωνώ με τον εισηγητή, δεν είναι καθόλου δημοκρατικό, διότι αρνούμεθα το δικαίωμα που έχει αυτή η Επιτροπή να ψηφίσει μια ολόκληρη σειρά τροπολογιών που αφορούν την ουσία του θέματος, δηλαδή κατά πόσο συστήνουμε ή όχι ε, να μην δοθεί σύμφωνη γνώμη και για διαδικαστικούς και δημοκρατικούς λόγους και για λόγους ουσίας είμαι κάθετα αντίθετη με αυτό και θα ήθελα να ζητήσω από το ΕΛΚ να πάει στην ψηφοφορία και να δεχθεί τα δημοκρατικά αποτελέσματα όπως εμείς και να μην προσπαθήσει να μην ψηφιστούν διάφορες βασικές τροπολογίες μέσω διαδικαστικών κόλπων. Από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ. Λέει και ο Σλίτα, συμφωνώ με την προλαλήσασα. Αλλά αν το ΕΛΚ συμπεραίνει ότι 37 είναι ασύμβατη, δεν έχει νόημα να ψηφίσουμε αυτήν πρώτα. Το μόνο λογικό συμπέρασμα θα ήταν να ψηφίσουμε συμβαστική 6 πρώτα, με απόφαση να απορριφθεί η άκτα, διότι συμβαστική 6 αφορά και την παράγραφο 9 και τη 15 και η συμβαστική πρέπει πρώτα να ψηφίζεται διότι είναι το πιο ευρύ συμπέρασμα είναι επίσης συμβιβαστική και καλύπτει και την παράγραφο 9, 9α. Όλα αυτά προηγούνται τις 37. Προτείνω να ψηφίσουμε συμβαστική 6 πρώτα και αν γίνει δεκτή η 37 καταπίπτει. Οπότε πάνε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Πρόεδρε, εν γέννη, λέει ο κύριος Κύρκοπ, δεν είναι θέμα πολιτικό. Ήταν λάθος αυτό που υπόθηκε. Τεχνικός πώς θα ευνοούσαμε τη θέση του ΕΛΚ και αυτά που είπαν όσον αφορά τη συγκεκριμένη τροπολογία. Αυτή είναι η θέση μας. Η Γκουε θα είμαι σύντομη, πάρα πολύ σύντομη. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι πιστεύω ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με αυτή την τεχνική λύση όπως παρουσιάζεται. Νομίζω ότι οποιοδήποτε είδε τον κατάλογο των ψηφοφοριών θα είχε διαπιστώσει αμέσως ότι υπάρχει σαφής πρόθεσης από πλευράς του ΕΛΚ να χρησιμοποιήσει την τεχνική διόρθωση για να αλλάξει την ουσία, το πρόσχημα αυτό. Η ΙΤΑ και οι Γιούρι καταψήφισαν την άκτα σήμερα. Πριν ψηφίσουμε θα πρέπει να σταθμίσουμε ακριβώς τι ψηφίζουμε. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε ασαφή αποτελέσματα. Λοιπόν, θέση της ομάδα μου είναι ότι θέλουμε κατάλογο ψηφοφοριών, ο οποίος είναι σαφής, ξεκάθαρος, που ταιριάζει με τον κατάλογο που πεστάλη χθε το βράδυ. Και ψηφίσαμε τη συμβαστική αν ψηφίσουμε την, καταψηφίσουμε τη συμβαστική έξι, τότε θα ακολουθήσουμε τη συνηθισμένη διαδικασία. Πρέπει να ακολουθήσουμε την κανονική διαδικασία. Διαφορετικά τελικά δεν θα εκπληρώσουμε το δημοκρατικό μας καθήκον. Νομίζω ότι κάποια πλειοψηφία είναι υπέρ του ισχύοντος καταλόγου ως έχει του καταλόγου ψηφοφοριών. Θα δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία στο ΕΛΚ να παρουσιάσει την προφορική του τροπολογία η ΔΕΜΗ θα πρέπει να απορρίψουμε χωρίς σχόλιο. Πρέπει να ψηφίσουμε τροπολογία 37 πρώτα και τα υπόλοιπα μετά. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με το πρώτο που είπατε. Να παραμείνει ο κατάλογος ως έχει, λέει ο κ. Μπουσετήλ. Διακόπτει ο Πρόεδρος είναι αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Όσον αφορά τις τροπολογίες και προσπαθούμε να αποφύγουμε τις συνέπειες. Δεν θέλουμε κάτι πάει στα 37 να καταπέσουν όλες αυτές που ακολουθούν. Η πρόταση του ΕΛΚ. Μετά την ψηφοφορία της 37, όλες οι σχετικές τροπολογίες που αφορούν το σχόλιο να καταπέσουν. Δεν το δεχόμαστε. Δεν υπάρχει συμφωνία με αυτή τη θέση. Η πλειοψηφία της Επιτροπής Λίμπε δεν το θέλει. Πρέπει να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες που σχετίζονται με την 97. Αυτή είναι η ερμηνεία της καταστάσεως. Yes, Simon. Please, let's not linger too much into it. Yeah, but Mr. Chairman, please allow me. This is a technical change. We were... Κύριε Πρόεδρε, αν με επιτρέπετε, είναι τεχνική αλλαγή ελέγχουμε τον κατάλογο ε, ψηφοφορίας όπως και όλες οι άλλες πολιτικές ομάδες. Οι πράσινοι, παραδείγματο χάρη, κάνουν, έχουν κάνει μάλλον ε, διάφορες προτάσεις ακόμη και μετά την υποβολή του δικού μας αιτήματος. Λοιπόν, εμάς είναι πολύ απλό αυτό που λέμε. Αν δύο τροπολογίες ουσιαστικά καλύπτουν το ίδιο πράγμα, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι συμβατέ μεταξύ του. Αν εγκριθεί η μία, καταπίπτει η άλλη εξού και σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να χρησιμοποιήσετε την εξουσία που έχει τός Πρόεδρος ε, και να αποφανθείτε από αυτού του τεχνικού αιτήματο. Αν η πλειοψηφία δεν θέλει τον κανόνα, δεν εφαρμόζει το κανόνας, δεν πάει έτσι το πράγμα. Αυτό το σύστημα ε, ανέκαθεν ισχύει και εφαρμόζεται στην Επιτροπή μας και όταν ε, υπάρχει μια τροπολογία που δεν είναι συμβατή με κάποια άλλη, πρέπει να καταπέπτει. Αυτό το κάνουμε ε, πανλημένως σε άλλες ψηφοφορίες. Σας παρακαλώ λοιπόν να φροντίσετε να τηρούνται οι κανόνες. Ο Πρόεδρος, το είπατε αυτό. Ακούσαμε όμως μετά ε, τις απόψεις και των άλλων πολιτικών ομάδων, γιατί το θέμα είναι τεχνικό. Και είναι και πολιτικό γιατί έχει να κάνει με τι επιπτώσει που θα έχει καταψήφιση τη τροπολογία 37 οι ομάδε θέλουν να ψηφιστούν οι υπόλοιπε ε, τροπολογίες που θα κατέπιπταν εάν ε, απερίπτω το 37. Και από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι λένε πρώτα να ψηφίσουμε το 37 και μετά τις υπόλοιπε. Ας ακούσουμε και τον κύριο Δρούτσα για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, διότι πραγματικά εργούμε για αυτό το διαδικαστικό θέμα και χάνουμε χρόνο. Κύριο Δρούτσα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω είπατε αυτό που έπρεπε. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι είναι λίγο απογοητευτικό ε, να βλέπει κανείς συναδέλφους από πολιτικές ομάδες να προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από ιονή διοικητικά θέματα και να συγκαλύψουν ένα άκρο πολιτικό ζήτημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε να πείτε ναι στην άκτα, κάντε το ανοιχτά, αγαπητοί συνάδελφοι. Μην προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από φυλάδια ή διοικητικά θέματα. There is issue involved. We should... Μα ακριβώς, ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε στην ψηφοφορία. Διαδικαστικό, κύριε Σλίτερ. Ακούστε, ο συντονιστής του ΕΛΚΑ έκανε άμεση αναφορά στους πρασίνους. Είπε ότι παίζουμε παιχνιδάκια. Εγώ υπέβαλα μια προφορική τροπολογία και να αρκεί ένα να σηκωθεί και να πει δεν τη θέλω αυτή την προφορική τροπολογία και αποσύρεται. Αυτή είναι η κανονική διαδικασία. Δεν είναι κανένα κόλπο. Μην με μπλέκετε στα βρώμικα σα παιχνίδια παρακαλώ. Well, that is okay. I think there is a majority to go on. Λοιπόν, όπω είπε ο κύριος Δρούτσας, λέει ο πρόεδρο, υπάρχει πλειοψηφία που λέει να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία και έτσι λοιπόν ξεκινάμε. Τροπολογία 1, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 με προφορική τροπολογία υπέρ Α, ναι, με συγχωρείτε, ο Άλβαρο. Επειδή είπε ε, ο κύριος Λίτερ ότι εάν κάποιο ε, τεθεί αντίθετο στην προφορική τροπολογία απορρίπτεται, εγώ ενίσταμαι, δεν δέχομαι την προφορική τροπολογία. Άρα πάει η προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε την αρχική τροπολογία 6. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 που είναι συμβατή με την 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Against. Abstention. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 καταπίπτει, καταπίπτει, καταπίπτει. Πάμε στην 9. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. 9 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Συγγνώμη. 9 πρώτο τμήμα υπέρ. 9 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 9 πρώτο τμήμα. Ελεκτρονικός έλεγχος. 9 πρώτο τμήμα. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 23-34 απορρίπτεται. Συμβαστική. Τρία, λέει ο πρόεδρος. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει, λέει ο πρόεδρος. Καταπίπτει, καταπίπτει. Τροπολογία 19. Listen, the second part of this amendment 9. Το δεύτερο τμήμα της 9 καλύπτεται από τη συμβαστική 3 που ψηφίσαμε μόλις τώρα. Είμαι σίγουρος. Εντάξει είμαστε. Πάμε στη 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 21. 21 έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Ένα σέλκ παραπάνω. Α, ενταξει πέρα ψηφοφορία. ψηφοφορίας. 23-34. Απορρίπτεται. 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ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 Αποχές εγκρίνεται. 32. Σε τρία τμήματα. Πρώτο, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 35 Α, 37 η διαβόητη τροπολογία 37 ας ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε τώρα σε 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε το κείμενο που τροποποιήθηκε τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Ένα μέλος του ΕΛΚ παραπάνω. Ένας ΕΛΚ παραπάνω. Μπορεί να κάνετε κάτι. Πέρας. Πέρας. 36 συν μια ψήφος μείων. Ευχαριστούμε κύριε Δρούτσα. Συγχαρητήρια. Στο. That'll be all. Εδώ ολοκληρώνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή, τη συνεργασία και την υπομονή. Τρεις το μεσημέρι ξανά εδώ. Γεια σας.